Bună ziua și bine ați venit la reuniunea comisiei noastre. Pentru prima parte a acestei reuniuni îmi uh, revine plăcerea. Αρχίζει η συνεδρίασή μας. Έχω την τιμή και την ευχαρίστηση να, προεδρε... να προεδρεύσω τη συζήτηση στο πρώτο τμήμα αυτή τη συνεδρίαση. γιατί ο πρόεδρο μα πρόεδρος μας έχει καθυστερήσει λίγο. Λοιπόν, το πρώτο σημείο τη ημερήσιας διάταξη είναι η έγκριση τη ημερήσιας διάταξη. Η ομάδα του ΕΛΚ ζήτησε να αποσυρθεί το σημείο 5. Προφορική ερώτηση με συζήτηση σχετικά με τις εισαγωγές βοήου κρέατος από τη Βραζιλία. Αυτό θα συζητηθεί στο πέρας της συνεδριασής μας. Επίσης σας πληροφορώ ότι το Συμβούλιο ζήτησε τη γνώμη του Κοινοβουλίου σε σχέση με μια νέα πρόταση της Κομισιόν σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού του για το γάλα, του, του ΠΟΗ για το γάλα και η Κομισιόν θέλει το θέμα αυτό να περάσει με τη διαδικασία επίγοντος. Προτείνω λοιπόν το σημείο αυτό να μπει στην ημερήσια διάταξη για ανταλλαγή απόψεων. Επίσης ε, συζητήθηκε για τη συνέχεια που θα δοθεί στις 19 Οκτωβρίου σε έκτακτη συνεδρίαση στο Στρασβούργο. Αν οι συνάδελφοι συμφωνούν, θεωρούμε ότι έχει εγκριθεί με αυτές τις αλλαγές η σε διάταξη. Σήμερα καλύπτονται όλες οι γλώσσες στη συνεδρίασή μας. Επίσης η συνδύασή μας ε, μεταδίδεται και μέσω διαδικτύου. Επόμενο σημείο, αηφόρος γεωργία και διατήρηση του εδάφους, το σημείο 3, το σχέδιο ΣΟΚΟ. Προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των γεωργικών μεθόδων και της διατήρησης του εδάφους, να αξιολογηθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο και οι πολιτικέ κινήτρων να αξιολογηθούν τα κενά του ισχύουσας Νομοθεσία και να δοθούν οι ιδέες πληροφορίες σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Καλωσορίζω τον κύριο Γκέι από το Ινστιτούτο της Σεβίλης και τον κύριο Μονταναρέλα από Ερευνητικό Ινστιτούτο της ΙΣΠΑ. Αυτοί θα μας παρουσιάζουν τα πορίσματα για την αηφόρο γεωργία και τη διατήρηση του εδάφους. Κύριε Γκέι, έχετε το λόγο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι ο Λούκα Μονταναρέλα και μαζί με τον συνάδελφό μου τον κύριο Γκέι θα παρουσιάσουμε στην Επιτροπή σας τα βασικά αποτελέσματα του ε, έργου αυτού. Ένα έργο δύο Ινστιτούτων του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Το ένα είναι στην Ίσπρα και είναι για το περιβάλλον και την ε, αηφορία και το άλλο είναι το Ινστιτούτο της Σεβίλης για τις προωθημένες τεχνολογικές έρευνες από όπου είναι ο κύριος Γκέι. Το πρώτο μέρος της παρουσίασης θα το κάνω εγώ και μετά θα δώσω τον λόγο στον Αλφο για τα συμπεράσματα. Το έργο αυτό στόχο έχει να αντιμετωπίσει την υποβάθμιση του εδάφους και τη γεωργία στην Ευρώπη, να σας δώσει μια γενική εικόνα για την κατάσταση όσον αφορά την υποβάθμιση του εδάφους γενικά στην Ευρώπη, καθώς και σχέση με διάφορες γεωργικές πρακτικές. Οπότε σύντομα θα παρουσιάσω την τωρινή κατάσταση στην Ευρώπη, όπως αυτή προέκυψε από τα αποτελέσματα του σχεδίου μας, καθώς και μια σύντομη επισκόπηση των ε, πρακτικών και στήματων που υπάρχουν για την διαφυλάξη του εδάφους. και μετά θα δώσω λόγο συνάδελφο για να σας πει τα βασικά στοιχεία ε, που προέκυψαν για το πώς θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι αγρότες της Ευρώπης για να υιοθετήσουν αηφόρες ε, πρακτικές. Ποια είναι τώρα λοιπόν η κατάσταση της υποβάθμισης του εδάφους στην Ευρώπη. Ε, σας την έχει παρουσιάσει ήδη η Κομισιόν το 2006 όταν ε, παρουσίασε μία ανακοίνωση προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο την ε, άποψή της για την θεματική στρατηγική προστασίας του εδάφους και βρήκαμε εκεί πέρα ποιες ήταν οι βασικές διαδικασίες ε, που λάμβαναν χώρα στην Ευρώπη όσον αφορά τα εδάφη και είχαν αυτό το αποτέλεσμα. Βέβαια δεν σχετίζονται αυτές όλες άμεσα με την γεωργία. Αυτές που σχετίζονται άμεσα είναι οπωσδήποτε η διάβρωση που είναι εκτεταμένη στην Ευρώπη και η διάβρωση από τον αέρα και από το νερό καθώς και η συνεχής μείωση του ε, του οργανικών υλών, η συμπίεση του εδάφους, αλλά και άλλες διαδικασίες που σχετίζονται με την γεωργία άμεσα ή έμεσα, όπως ε, παραδείγματο χάρη η αλάτωση και η οξύνηση σε κάποια σημεία την Ευρώπη. Επίσης ε, το ότι υπάρχει σφράγιση θέλετε, του εδάφους λόγω κατασκευών, κατοικίας κτλ. καθώς και μόλυνση τοπική και γενικότερη και τέλος κατολιστήσεις που συχνά επίσης προκαλούν ε, απώλειες μέχρι και ανθρώπινων ε, ζώων. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ε, το έργο αυτό, το σόκο το λεγόμενο, επικεντρώθηκε κυρίως στι στις διαδικασίες οι οποίες έχουν σχέση με τη γεωργία, δηλαδή η διάβρωση, συμπίεση, μείωση των οργανικών υλών, αλάτωση και οξύνηση. Πρώτα απ' όλα λοιπόν η απογύμνωση του εδάφους δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχουν κάποιες ε, περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο, άλλες ε, λιγότερο, οπότε πρέπει να τις δούμε σε ένα χάρτη. Εμείς έχουμε αρκετούς θεματικούς χάρτες που τονίζουν αυτές τις διαδικασίες. Βλέπετε εδώ πέρα το χάρτη της διάβρωσης όπου βλέπετε τις περιοχές όπου, που κινδυνεύουν περισσότερο από διάβρωση από νερό. Τα πιο κόκκινα χρώματα βλέπετε ότι είναι πιο κοντά στην Μεσόγειο, είναι οι περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο. Επίσης αξιολογήσαμε την ε, τωρινή κατάσταση του οργανικού άνθρακα και του ποσοστό του ποσοστού του στα πρώτα 20 εκατοστά των γεωργικών γεών και όπως βλέπετε υπάρχει μια σαφή τάση πάλι βορρά-νότου. Παραδοσιακά όπως ξέρετε σε πιο κρύα και ψυχρά περιβάλλοντα έχουμε υψηλότερο ποσοστό στο έδαφος. Οπότε υπάρχει υψηλό ποσοστό στη Βόρεια Ευρώπη και χαμηλότερο στη Νότια Ευρώπη. Αλλά αυτό το οποίο ήταν πιο ενδιαφέρον οπωσδήποτε ήταν οι άλλες διαδικασίες ε, όπως ξέρετε, υπολογίζεται ότι έχουμε 70 γιγατόνους αποθηκευμένους σε οργανικό άνθρακα σε αυτή την κατάσταση. Γνωρίζουμε λοιπόν πως είναι μια δυναμική ισορροπία στα εδάφη. Αν δείτε αυτό το γράφημα έχουμε το αποτέλεσμα όταν ξεκινάμε δηλαδή από μια ονομαστική κλίμακα του 100 ε, πριν τη μετατροπή χρήσης ε, γης, δηλαδή πριν ξεκινήσουν να παράγουν σε ένα σταθερό επίπεδο τα εδάφη. Όταν ξεκινήσουμε λοιπόν την γεωργία, κατά κανόνα έχουμε και αύξηση των μεταλλικών ε, στοιχείων και φτάνουμε σε ένα νέο σημείο ισορροπίας που ανάλογα με τα νέα συστήματα γεωργίας είναι λίγο πολύ σταθερό εκτός εάν υπάρχει μια επιταχυμένη διαδικασία Διάβρωση Στόχος ήταν να δούμε ποιες τεχνικές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να προτείνουμε ε, τεχνικές που χρησιμοποιούνται ήδη σε κάποια μέλη της Ευρώπης για να επαναφέρουμε στα υψηλότερα επίπεδα τον οργανικό άνθρακα με φόρους πρακτικές για να φτάσει και στο ιδανικό επίπεδο που είναι το φυσικό και σταθερό αλλά μπορούμε να πάμε και πάνω από το ε, επίπεδο αυτό. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι πρακτικές που εξετάσαμε. Κατ' ουσίαν εξετάσαμε δύο συστήματα, το σύστημα ε, διατήρησης, ε, συντήρησης, ένα σύστημα στο οποίο γίνεται μειωμένη ή και καθόλου ε, άρρωση, οπότε εκεί πέρα δεν υπάρχει αυτή η αποψήλωση του οργανικού άνθρακα. Συχνά αυτό το σύστημα μειωμένης ε, καθόλου άρρωσης ε, γίνεται σε συνδυασμό με άμυψη σπορά. Το άλλο το οποίο είδαμε είναι η βιολογική γεωργία που οπωσδήποτε γνωρίζετε καλά. Κατόπιν υπάρχουν κάποιες πρακτικές γεωργικές ε, όπως π.χ. προστατευτικές καλλιέργειες, άμυψη σπορά, εμβόλυμη καλλιέργεια, καλλιέργεια στις ράχες, υπεδάφιος άρρωση, καλλιέργεια κατά τις υψοϊψής καμπύλες, όλα αυτά δηλαδή τα οποία ευνοούν τη διατήρηση του εδάφους, επίσης λουριά, αναβαθμίδες και αλλαγές χρήσης γης όπως π.χ. αγροδοσοκομεία ή χορτολιβαδικές εκτάσεις. Όλα αυτά βεβαίως έχουν πλεονεκτήματα και από ε, περιβαλλοντική και από οικονομική πλευρά, όπως και μειονεκτήματα. Τα συστήματα ε, γεωργίας τα οποία είδαμε είναι αυτό το οποίο κατά βάση σας είπα είναι η λεγόμενη γεωργία προστασίας διατήρησης, δηλαδή υπάρχει ενσωματωμένη σε αυτήν η προστασία του εδάφους και μειώνεται έτσι η αποψήλωση του οργανικού άνθρακα από το και η διάβρωση του εδάφους, αλλά μπορούμε να έχουμε και υψηλέ αποδόσεις. Η βιολογική γεωργία εξετάστηκε όσον αφορά τα πλεονεκτήματα στην ε, μείωση της μόλυνσης του εδάφους καθώς ε, δεν χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες, ενισχύεται η βιοπικιλότητα, υπάρχει επίσης ε, ένταξη σε μια συγκεκριμένη πλευρά της αγοράς, αλλά βεβαίως από την άλλη μεριά υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος στην στρεματική απόδοση. διαφορετικές προσεγγίσεις οι οποίες όμως έχουν και οι δύο προβληματικές στοιχείες, δηλαδή πρόκειται για περίπλοκα στήματα που απαιτούν μια, ένα αρκετά μεγάλο βαθμό τεχνολογικής εξειδίκευσης. Υπάρχει μεγάλο κόστος για να γίνει μετατροπή, κόστος και σε γνώση και σε εξοπλισμό. Είναι μεγάλη περίοδος της προσαρμογής και χρειάζεται να υπάρξει και μια προσαρμογή σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες, περιβαλλοντικές συνθήκες Ευρώπης. Οπότε είδαμε και την αποτελεσματικότητα αυτών των μετατροπών, αυτά τα οποία παρατηρήσαμε σε πολλές από τις πιλωτικές εκτάσεις που είδαμε. Οι φάσεις λοιπόν αλλαγής και μετατροπής, π.χ. για να πάμε σε μια καλλιέργεια προστασίας, συχνά στην πρώτη φάση έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής και του κέρδους του αγρότη, που μπορεί να είναι βεβαίω αυτός ένας από τους λόγους για τους οποίους οι τεχνολογίες δεν υιοθετήθηκαν σε κάποια μέρη της Ευρώπης. Οπωσδήποτε μακροπρόθεσμα παρατηρούμε πως υπάρχει αύξηση της ε, παραγωγής για την ε, γεωργία αυτή της ε, προστασίας και αυξάνεται το ποσοστό στο γενικότερο σύνολο της γεωργίας. Όπως σας είπα δεν μπορούμε να δούμε τώρα όλες τις λεπτομέρειες. Έχουμε όπως σας είπα στοιχεία πάρα πολύ αναλυτικά για όλες αυτές τις πρακτικές, προστατευτικές καλλιέργειες, άμψης φορά, ευόλυμες καλλιέργειες, καλλιέργεια κατά τη ισοϊψής και για το αποτέλεσμα το οποίο είχαν κάποιες από αυτές τις πρακτικές οπωσδήποτε είναι πρακτικές οι οποίες παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν, π.χ. αναβαθμίδες χρησιμοποιούνται παραδοσιακά ε, στη Μεσόγειο, αλλά και άλλα συστήματα καλλιέργειας. Καταλήγοντας λοιπόν στο πρώτο τμήμα της ε, παρουσίασης, τα αποτελέσματα έδειξαν οπωσδήποτε πως υπάρχουν πολλές τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους αγρότες για να αυξηθεί η προστασία. Υπάρχουν και άλλες τεχνικές τις οποίες δεν εξετάσαμε. Κάθε μία από αυτές ε, τις τεχνικές έχει θετικές και αρνητικές πτυχές. Οπωσδήποτε θα πρέπει να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες συνθήκες και εδάφους και υδάτων. Οπότε δεν υπάρχει μία συνταγή για ολόκληρη την Ευρώπη. Πρέπει να υπάρχει τοπική προσαρμογή. Ειδικά τώρα για το ζήτημα της γεωργίας αυτής της προστασίας Μα έδειξαν τα αποτελέσματα πως είναι υποσχόμενη τεχνολογία, αλλά σημαίνει πω απαιτούνται πολύ σοβαρέ αρχικέ επενδύσει, εξειδικευμένη γνώμη και λεπτέ παρεμβάσει για να αποφευθεί η χρήση χημικών και να μην υπάρξει μείωση της θερματική απόδοση. και τέλο, όπω σα είπα χρειάζονται ε, αρκετά μακροχρόνιε περίοδοι προσαρμογή μέχρι να φτάσουμε σε κάποια ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τέλο, θα δώσω στην συνάδελφο για να περάσει τα συμπεράσματα. Θα δώσω λόγο στην άλφα. Um, uh, um, Συνεχίζοντας, εξετάσαμε το περιβάλλον από πλευράς πολιτικής και, σε κάθε βελτίωση που εξετάζουμε πρέπει να δούμε ακριβώς που εντοπίζεται, οπότε θα πρέπει να υπάρχει κάποιο σημείο αναφοράς. Οπότε θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το επίπεδο αναφοράς και αυτό το επίπεδο αναφορά θα πρέπει να είναι υποχρεωτική ρύθμιση, αλλά θα πρέπει να βελτιωθεί. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει κάποιο στόχο ε, υψηλότερο. Και αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στα μέτρα που λαμβάνει κανεί. Οπότε το επίπεδο αναφορά θα πρέπει να αφορά αυτά τα υποχρεωτικά μέτρα, κάτι που να τηρίζουν όλοι και παραπέρα. Θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια κίνητρα όσον αφορά κάποιε πληρωμέ. ή τέλο πάντων να υπάρχει περισσότερη συνειδητοποίηση, οπότε θα πρέπει να υπάρχει και ενημέρωση του κόσμου για τι δυνατότητε που προσφέρονται. Το α, πλαίσιο αυτό, εδώ σα αναφέρω τι με, με τι ε, ε, πολιτικέ και τώρα μπορείτε να δείτε τι γίνεται στα πλαίσια τη ΚΑΠ και βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουμε βέβαια εδώ πέρα ε, την πολλαπλή συμμόρφωση μεταξύ των άλλων γιατί έχουμε και νομοθεσία από άλλες πολιτικές που θα πρέπει και αυτή να ενσωματωθεί και να τηρηθεί ε, σε σχέση με την πολλαπλή συμμόρφωση. Θα πρέπει να τηρούνται πάντοτε και οι διατάξεις που βοηθούν το περιβάλλον, κάποιες ρυθμίσεις που αφορούν την προστασία του εδάφους και όλα αυτά αναφέρονται σαφώς ε, όσον αφορά κάποιες ουσίες ε, ε, κάποιες ουσίες οργανικές οπότε υπάρχουν αυτά τα μέτρα τα οποία αφορούν το περιβάλλον και φτάνουν μέχρι εκεί που να τηρούνται κατευθύνσεις που έχουμε δώσει προς τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Βλέπετε εδώ πέρα τώρα ποιο είναι το, ποια είναι η πολιτική για το περιβάλλον και Βλέπετε εδώ αυτά τα τετραγωνάκια που έχουμε χρωματίσει με ανοιχτό μπλε και αναφέρονται τα νομοθετήματα που σχετίζουν με την κοινή αγροτική πολιτική ε, και την προστασία του εδάφους και τώρα όλα μαζί το βλέπετε πάνω πάνω έχουμε κάποιους στόχους όπως ας πούμε την διάβρωση από το νερό. Εδώ βλέπετε κάποια συστήματα, κάποιες πρακτικές που ακολουθούνται και εξετάζονται. Ε, βλέπετε ποιες πολιτικές βοηθούνται. Ε, και ανάλογα με το πόσο έχουν σχέση με κάποια πολιτική, με κάποιο μέτρο είναι το τετραγωνάκι άσπρο, ή κίτρινο ή πράσινο όταν είναι, ε, κάτι το οποίο βοηθά το, την πολιτική του το περιβάλλον. Ούτως ώστε με κάποιες πολιτικές να ενθαρρύνονται οι ε, αγρότες να κινηθούν προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τώρα, ρίξτε μια ματιά στο τι γίνεται σε τοπικό επίπεδο που είναι πολύ σημαντικό. Να δείτε πώς εφαρμόζεται το κάθε μέτρο Έχουμε κάνει κάποιες στοχευμένες με μελέτες. Σε Δύση, Νότο, σε όλη την Ευρώπη γενικά και είδαμε ότι ξέρουν ποιες είναι οι προκλήσεις οι Γεωργοί. Και όσον αφορά την προστασία του εδάφους, δεν θεωρούν ότι τα πράγματα πιέζουν τόσο πολύ. Ξέρουν ότι πρόκειται για κάποια πρόκληση, αλλά δεν θεωρούν ότι είναι κάτι που πρέπει να του απασχολεί καθημερινά. Και τελικά συνεχίζουν να κάνουν ό,τι κάνουν συνήθω μέχρι ότου δουν κάποιε συνέπειε στην εκμετάλλευσή του. Πολλέ φορέ δεν έχουν αρκετή ενημέρωση και πληροφορίε, οπότε έτσι εμποδίζεται η εφαρμογή νέων μέτρων που θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ ωφέλιμα. Επίσης, πολλές από τα πράγματα είναι ανάμεικτα, δηλαδή αλλού υπάρχουν κάποια κίνητρα, αλλού υπάρχει υποχρεωτικό της εφαρμογής. Οπότε, από εκεί ξέρετε το κατά πώς να εφαρμοστεί ένα μέτρο. Από το να ξέρει ο άλλος πώς θα ενεργήσει. Και χρειάζεται τώρα κάποια αξιολόγηση για το ποιε είναι οι επιπτώσει κάποια πολιτική όσον αφορά την πρόσταση του εδάφου. Μια που τα πράγματα είναι τόσο περίπλοκα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί ποια είναι η τελική συνέπεια μια πολιτική σε ενωσιακό επίπεδο. Απλό προστασία του εδάφου. Είναι δύσκολο να βρεθεί ότι ο Τώρα όμως βλέπουμε όλο το ψηφιδωτό μαζί και βλέπουμε για κάποια μέτρα τα οποία ε, διατίθενται, τα οποία υπάρχουν, τα οποία προβλέπονται. Βλέπουμε επίσης ε, κάποια να είναι πιο πρόσφορα από άλλα. Και είδατε ότι η υπολοπλή συμμόρφωση βοήθησε να υπάρχει τελικά ένα κοινό επίπεδο αναφοράς. Βλέπετε επομένως εδώ τι είναι υποχρεωτικό να γίνει από όλους, βασικό επίπεδο, ε, ποιο θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος κοινός παρονομαστή, το ελάχιστο του των τηρουμένων. Βλέπουμε ότι πάρα πολύ σημαντικό τμήμα της όλης πορείας είναι το μεταβατικό στάδιο. Δηλαδή η μετάβαση από το ένα σύστημα στο Άλλο από τη μία πρακτική στην άλλη. Εδώ παίζει μεγάλο ρόλο, πολύ σημαντικό ρόλο η πληροφόρηση. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συντονισμός. Συντονισμός και με άλλες πολιτικές, άλλα μέτρα που έχουν στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς θα γίνει η διάδοση αυτής της ιδέας. Ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή την ιστορία. Και κατόπιν προχωρήσαμε σε έρευνα. Συγκροτήθηκαν κάποια εργαστήρια, ένα σεμινάριο χάραξης πολιτικής Έχουμε όλες τις εκθέσεις που έχουν συνταγή, ε, δύο είναι οι πιο βασικές από αυτές και τις δύο μπορείτε να τις βρείτε στο website ε, και ξέρετε τις, τις έχουν κατεβάσει αυτές μέσα για να διαβάσουν 15.000 φορές. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πόσα πέρασαν τα εργαστήρια κλπ. Έχουμε αυτά τα ενημερωτικά δελτία, fact sheets, σε πάρα πολλές γλώσσες τα έχουν μεταφράσει. Η ε, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία έχουν ενδιαφερθεί πάρα πολύ και έχουν κατεβάσει τι αντίστοιχε μεταφράσει. Βλέπετε εδώ πέρα τι άλλο υπάρχει από αυτά τα ενημερωτικά φυλάδια, τι άλλο υπάρχει στο Ιντερνετ. Τέσσερι σελίδε. Ένα θέμα, Βλέπετε εδώ πέρα αυτές τις όλες ιδέες στα διάφορα επιμερισμήματα. Ε, εδώ τελειώσαμε. Σας ευχαριστούμε. Λεφόλ, ha chiesto Στεφάν, excuse me. έχετε το λόγο. Στεφάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όμω, θα πρέπει πρώτα πρώτα να ευχαριστούμε του δύο εκπροσώπου τη Κομισιόν. Μα παρουσίασε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο όντω ε, ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Κατρίν Κικέ και ο υποφαινόμενο. Το ξεκίνησαμε αυτό και θελήσαμε να έρθουμε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε να υπάρξει μια αξιολόγηση, να υπάρξει μια καταγραφή εκ νέου των ε, γεωργικών πρακτικών σε όλη την Ευρώπη. Και το πιο βασικό το οποίο ακούσαμε ήταν το, το σχετικό με την προστασία του εδάφου. Γιατί στην Ευρώπη, όπω και παντού, προχωράει η διάβρωση του εδάφου. Και ανέφερε στου αδέλφου ότι θα πρέπει να μην ξεχνάτε ότι όσον αφορά το σύνολο τη γη, το σύνολο υδρογείου, το έδαφο του οποίου ε, έχουμε την παραγωγή, την, την γεωργική, ε, έχει μειωθεί κατά 30 εκατοστά. Ε, ή μάλλον συγγνώμη, ότι η Γεωργία ασχολείται και διαχειρίζεται 30 εκατοστά από όλη αυτή την σχετική επιφάνεια. Επομένω, η προστασία του εδάφου είναι μια πάρα πολύ σημαντική διάσταση, είναι κάτι το οποίο μας περιορίζει, είναι τη της μας, κάτι το οποίο έχει εξηγηθεί και στο βορρά και στο νότο της Ευρώπης, γιατί έχουμε διάφορου τύπου ε, απομείωσης, ε, το κρύο, η ζέστη υγρασία και οι τεχνικές παραγωγές, οι γεωργικές που και αυτές οι ίδιες έχουν επιφέρει την ε, απομείωση του εδάφους. Άρα θα πρέπει να γίνει μια σφαιρική ανάλυση του, του, του παράγοντα του κλιματικού, ποιες είναι οι συνέπειες επί του εδάφους, οπότε θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι είναι προς το συμφέρον μας να προστατεύσουμε το έδαφος, και επίση θα πρέπει να δούμε ότι το έδαφος έχει την ιδιότητα να κατακρατεί να, τις οργανικές ουσίες και τον άνθρακα. Σήμερα έχουμε 70, δισεκατομμύρια δις εκατομμύρια τόνων άνθρακα που κατακρατούνται από το έδαφος. Δύο δις ε, κατά μέσο όρο ε, πετάμε στην Ευρώπη. Οπότε μπορεί να καταλάβετε ποια είναι η σχέση αυτού του στοιχείου με την ε, άνοδο της του πλανήτη. Επομένως, αυτό το πρόγραμμα ξεκινά με το πώς θα φρενάρουμε την απομείωση του εδάφους. Γίνεται μια καταγραφή των τεχνικών που θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε το στόχο μας και τα δύο στοιχεία τα οποία τονίστηκαν είναι η βιολογική γεωργία γιατί λένε οργανική και από την άλλη έχουμε κάποιες νέες τεχνικές, τις τεχνικές προστασίας, διατήρησης του εδάφους. Και αυτό που πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι όταν μιλούμε για προστασία του εδάφους έχουμε αυτές τις τεχνικές που μας οδηγούν σε κάποια νέα μοντέλα παραγωγής Ούτω ώστε με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο να μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση στο ερώτημα του πώς θα διαμορφώσουμε την βιώσιμη γεωργία του αύριο Ούτω ώστε να δούμε πώς θα είναι και παραγωγική και αποδοτική η γεωργία και ταυτόχρονα να είναι ε, υπεύθυνοι οικολογικά. Συζητάμε εδώ πέρα για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Όλο το κοινοβούλιο ασχολείται με αυτό και θέλουμε να λάβει υπόψη η γεωργία των παράγοντα περιβάλλον. Όμως τώρα θα πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στα έργα. Να δώσουμε κάποιες απαντήσεις συγκεκριμένε στους γεωργούς, οι οποίοι όπως ελέγχθη ξέρουν ποιες είναι οι προκλήσει που έχουν αντιμετωπίσουν. Οπότε, με αυτή την λογική, με αυτό το πνεύμα τη ε, προστασία του εδάφου έχουμε διαμόρφωση του αυριανού μοντέλου παραγωγή που θα είναι και παραγωγικό και θα είναι και οικολογικά υπεύθυνο, κάτι το οποίο μας το δείχνουν αυτές οι καμπύλες, αυτά τα γραφήματα τα οποία τα είδαμε στην παρουσίαση ούτω ώστε να μπορέσουμε τελικά με τις νέες τεχνικές να έχουμε και την παραγωγή που εξασφαλίζει η παραδοσιακή γεωργία, αλλά και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να έχουμε βιώσιμη γεωργία και να προστατεύσουμε το έδαφο και κλείνω με ένα στοιχείο το οποίο σα προσθέτω ότι μιλούμε για την προστασία του εδάφου με κάποιε τεχνικέ οι οποίες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσε και για άλλους στόχου. και οπότε στο μέλλον θα πρέπει στο Κοινοβούλιο αλλά και στην Κομισιόν να συζητούμε για την γεωργία σε σχέση με το περιβάλλον με τρόπο σφαιρικό. Να σταματήσουμε ζητούμε να έχουμε επιμέρους ε, αντιμετώπιση, οδηγία για τα ύδατα, για τα ε, φυτοφάρμακα κλπ. Θα πρέπει τα μέτρα να είναι εγκάρσια, να είναι συνολικά όπως είναι και το πρόβλημα τέτοιο. Και μόνο έτσι θα καταλήξουμε σε κάποιες λύσεις. Αυτό είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζει αυτό το project που παρουσιάστηκε και έτσι να μπορούμε να φτάσουμε σε μια τεχνοκρατική σύντηση για το μοντέλο παραγωγής. Αυτό ήθελα να σας πω που είναι το πιο σημαντικό. Βρισκόμαστε στην πρώτη φάση της διαδρομής. Σας ευχαριστούμε για το έργο που επιτελέσατε. Είναι εξαιρετικό. Είναι σωστά είναι σωστή η σύλληψή του και ε, έτσι μπορεί να μας δείχνετε πώς είναι τα πράγματα σε μια προοπτική ούτως ώστε να μπορέσουμε να βρούμε απάντηση για το ερώτημα του πώς θα πετύχουμε η γεωργία και να μπορεί να θρέψει τον κόσμο και ταυτόχρονα να είναι βιώσιμη. Αυτό ήθελα να σας πω και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους όσοι δούλεψαν για αυτό το project, το πρόγραμμα. Σε ευχαριστούμε Στεφάν. Πάρα πολύ σημαντικό το θέμα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Μάρτιν Χόσλινγκ έχει το λόγο τώρα. Να ευχαριστήσω και εγώ την Κομισιόν και βλέπετε πόσο επίγον είναι το θέμα από τους χάρτες. Είναι πολύ συγκεκριμένος ο κίνδυνος, η πιθανότητα κινδύνου και πρέπει να τα ξαναδεί αυτά το κοινοβούλιο γιατί έχει μπλοκαριστεί η προστασία του εδάφους σε πολλές περιπτώσεις αλλά πρέπει να ξαναμπεί στην ημερήσια διάταξη είναι πολύ πιο επίγουσα από ποτέ γιατί θα επιδεινωθεί και με την κλιματική αλλαγή. Και εμείς οπωσδήποτε θα το θέσουμε στην ημερήσια διάταξη. Έχω όμως ερωτήσεις γιατί τα είπατε πολύ γρήγορα. Είπατε πως η... μία προσέγγιση θα είναι η ε, ελάχιστη καλλιέργεια. Ίσως, αλλά με αυτό τον τρόπο υπάρχει πολύ έντονη χρήση χημικών ε, ουσιών και δεν ξέρω εάν ε, αυτό είναι σωστό ως αποτέλεσμα, δηλαδή να οδηγηθούμε στην ολοκληρωτική χρήση ζανιοκτώνων και κάνουμε ζημιά απλά προς μία άλλη κατεύθυνση. Είπατε σωστά πως η βιολογική γεωργία λόγω της ε, προσέγγισης της θα μπορούσε να αποτελέσει μία απάντηση πράγματι θα μπορούσαμε να προωθήσουμε τη βιολογική γεωργία. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει συγκεκριμένα και δυστυχώ δεν είπατε νούμερα είναι η περαιτέρω εντατικοποίηση της ε, γεωργίας και ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, παραγωγή γάλακτος καθώς χρειάζονται όλο και περισσότεροι βοσκότοποι και βλέπουμε πως ε, χρειαζόμαστε χορδολιβαδικές εκτάσεις γιατί αυτές εμποδίζουν και την διάβρωση αλλά βλέπετε πως ε, συνεχώς χορδολιβαδικές εκτάσεις καλλιεργούνται για να καλλιεργηθεί καλαμπόκι για ζωοτροφές. Πρέπει να το δούμε αυτό κάπως κεντρικά και μετά είπατε πολλαπλή συμμόρφωση μπορεί να αποτελέσει μια εγγύηση για τις σωστές πρακτικές. Κατά την άποψή μου οι τωρινές διατάξεις πολλαπλής συμμόρφωσης δεν επαρκούν, πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε γιατί ήρθα λίγο αργά. Οπότε δεν άκουσα τις παρουσιάσεις, αλλά τα ξέρω. Τα θέματα, έχει δίκιο συνάλφος, είναι σημαντικά τα ζητήματα. Θα ήθελα εγώ, κύριε, πρόεδρε, κύριε συνάλφε εδώ πέρα, να σας παρακαλέσω να προσέξετε. Μην τα κάνουμε όλα μαζί πακέτο. Έχουμε άνω των 300 τύπων εδαφών στην Ευρώπη και η κατάσταση διαφέρει πάρα πολύ στην Ευρώπη. Γνωρίζω μια μελέτη του ΟΗΕ, νομίζω στα μέσα της δεκαετίας του 90, που ερευνήθηκε παγκοσμίω που είναι η μεγαλύτερη ζημία του εδάφους. Και εκεί πέρα η Ευρώπη έχει τη μικρότερη ζημία του εδάφους. Είναι η Κεντρική και η Νότια Αμερική η μεγαλύτερη καταστροφή του εδάφους και αυτό σχετίζεται με τις γεωργικές δομές. Γιατί εκεί που υπάρχουν μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις και καλλιεργούν τεράστιες εκτάσεις με, φυτίε με φυτίες Εκεί λοιπόν αυτές οι μεγάλες ε, εταιρείε δεν δίνουν καμία βάση σε τίποτα παρά μόνο στα κέρδη τους. Οι δικοί μου αγρότες τώρα στη δική μου περιοχή που εργάζονται πηγενιές στην ίδια γη και θέλουν στην επόμενη γενιά, δηλαδή στα παιδιά τους να παραδώσουν η γη, γη εκεί πέρα προσέχουν το έδαφος και υπάρχει αηφόρος καλλιέργεια, οπότε πρέπει να προσέξουμε να υπάρξει αυτή η αηφόρος καλλιέργεια. Σήμερα έχουμε καλές δυνατότητες και νομίζω μπορούμε να διατηρήσουμε την ε, αηφορία του εδάφους. Αν δούμε σήμερα αυτά τα τεράστια τρακτέρ με τα τεράστια ελευνικούμενα πίσω και τα λάστιχα τα μεγάλα έχουν ελάχιστη πίεση την οποία ασκούν στο έδαφος. Οπότε Θέλω εδώ πέρα να σας προειδοποιήσω, δεν υπάρχει λόγος να δημιουργήσουμε νέα γραφειοκρατία στην Ευρώπη και να θεωρούμε πως με διατάξει στην Ευρώπη, στην, από τις Βρυξέλλες, μπορούμε να ρυθμίσουμε κάθε περίπτωση. Είναι πάρα πολύ διαφορετικές περιστάσεις μεταξύ τους και δεν είναι θέμα ευρωπαϊκό το έδαφος, είναι εθνική υπόθεση των 27 κρατών μελών μέσω της ανάλογης εθνικής νομοθεσίας να φροντίσουν ότι προστατεύεται το έδαφος στην χώρα τους και εγώ δεν θέλω πάλι από τις Βρυξέλλες να δημιουργήσουμε καινούρια ε, γραφειοκρατία, το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν, ορίζουμε νέες ε, ημερομηνίες ε, γιατί λέμε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξέρω εγώ, το τάδε προϊόν μέχρι τέλος ε, Φεβρουαρίου και μπορεί να είναι πιο συμφέρον να αγοραστεί κάτι μέχρι ε, ξέρω εγώ, αρχές Μαρτίου. Δεν είναι δυνατόν να ορίζουμε εδώ πέρα από τις Βρυξέλλες την τελευταία λεπτομέρεια και να δημιουργούμε νέα γραφειοκρατία συνεχώς. E Κι εγώ είχα μια και εγώ ζητάω συγγνώμη. Ζωζέ Καταρχήν ευχαριστώ και εγώ για την ε, δουλειά που έκανε ο Στεφάλε Φόλ με την ομάδα της Κομισιόν. Θα επανέλθω σε μια βασική αρχή που δεν αναφέρθηκε στην αρχή, που τη θεωρώ όμω δεδομένη. Το έδαφος δεν είναι ένα υπόστρωμα, είναι κάτι το ζωντανό. Από τη στιγμή που μιλάμε για το έδαφος, όχι σαν ένα υποστήριγμα αλλά σε ένα πολύπλοκο ζωντανό οργανισμό, τότε η καλλιέργεια της γης είναι διαφορετική έννοια. Πρέπει να το πούμε αυτό από την αρχή. Δύο παραδείγματα. Ανδαλουσία, είδαμε το πρόβλημα πως τίθεται από μια γεωργία με θερμοκήπια εντατική με ένα σωρό προβλήματα, αζωτούχα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κλπ. ή ένα γαλλικό πρόβλημα, η μονοκαλλιέργεια των σιτηρών. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα στήρωσης κυριολεκτικά του εδάφους, γιατί δεν ενσωματώνεται η μονοκαλλιεργεια των σιτηρων και αυτο ειναι ενα προβλημα στήρωση κυριολεκτικα του εδαφους γιατι δεν ενσωματωνεται η αρχη της αμυψης σποράς κλπ. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό θα μπορούσαμε ενδεχομένω να προβάλλουμε νέα σχήματα καθολικά, όχι γραφειοκρατικά, σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινή πολιτική. Δηλαδή, ξεκινήσαμε το 57 με μία κάπ με στόχο να αυξηθεί η παραγωγή για να τραφεί ο πληθυσμό της Υπήρου και ο καταναλωτή να έχει φτηνά τρόφιμα. Τώρα πρέπει να βάλουμε και νέα σχήματα στην καλλιέργεια και σε σχέση με το περιβάλλον. Σε δύο μήνες έχουμε την Κοπεχάγη. Η Επιτροπή Γεωργίας θα μπορούσε να επιλέξει ένα καινοτόμο τίτλο και να πει για τη Γεωργία ένα νέο αγροτικό πρόγραμμα θα επιτρέψει να ψυχρανθεί ο πλανήτης. Θα μπορούσε αυτός να είναι το αντικείμενο μιας νέας ΚΑΠ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε Ζωζέ. Ο κύριος Νταντά. Ευχαριστώ τους όσους μίλησαν για την πολύ ωραίες εισηγήσεις τους. Εδώ και 50 χρόνια η ανάπτυξη της γεωργίας κάπως ε, αποσχίστηκε από το θέμα της γεωπονίας. Γιατί, διότι η γεωπονία υποχώρησε στην έρευνα. Η γεωπονική υποχώρησε σε όλες τις μορφές γεωργικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πρέπει να κάνουμε σοβαρή δουλειά εδώ στην Επιτροπή έτσι ώστε η επιστήμη του εδάφους να ξαναπροβληθεί. Είναι μια καθολική επιστήμη και ο προηγούμενος ο Στεφάν Λεφόλ ο μιλητής είπε ότι πρέπει να έχουμε κατακόρυφες οδηγίες. Χρειαζόμαστε όμως και οριζόντιες πράξεις. Γιατί η αλήθεια για το έδαφος σε κάποιο τομέα δεν είναι ίδια με ό,τι ισχύει σε έναν άλλο τομέα. Συμφωνώ με τον Στάφο Μπερντές ως προς το ότι θα μπορούσε αυτό να το επισημάνουμε στο Συμβούλιο και δεν μιλάω για το Οικονομικό Συμβούλιο μόνο για τις ενισχύσεις γιατί το μέλλον της γεωπονικής και της καλλιέργειας του εδάφους είναι κάτι που αφορά το μέλλον όλων μας. Πρόεδρος, Τζον Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ενδιαφέρουσα μελέτη, αλλά δεν συμφωνώ ότι αυτό θα έπρεπε να μπει ε, στα πλαίσια της ε, ε εγκάρσιας ε, συμμόρφωσης, cross compliance. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ρυθμίζεται αυτό. Αν κάποιος επιτρέψει το έδαφος του να χειροτερέψει, μπορεί ο ιδιοκτήτης της γης να τον διώξει από τη γη αυτή, ένας το χάρη αν επιτρέψει ένας γεωργός το χώμα να βγει στην δημόσια εδώ, το, το, κοινοτικό συμβούλιο θα πάρει μέτρα εναντίον του. Ένας ιδιοκτήτης της γης, ένας ο οποίος κατέχει γη, θέλει να κρατάει τη γη του σε καλή κατάσταση. Πρέπει να διατηρεί την κεφαλογική αξία του αγαθού αυτού. Δεν θα το επιτρέψει σε καμία περίπτωση από μόνο του να χειροτερέψει. Μιλάμε για οργανικά υλικά. Νομίζω ότι αυτός δεν είναι καλός δείκτης για την υγεία του εδάφους. Μερικά εδάφη έχουν ψηλό οργανικό δείκτη, αλλά δεν συμβαίνει αυτό παντού, γιατί μπορεί να υποστούν έντονη διάβρωση. Η, οργανική ύλη δεν τους βοηθάει. Δεν υπάρχει εγγύηση δηλαδή για την οργανική ύλη σε κάθε Μερικά από τα πιο παραγωγικά εδάφη μα είναι χαμηλά σε οργανική ύλη. Και αν πάμε να αυξήσουμε την οργανική ύλη, παραδείγματος, χάρη δεν κάψετε την, της, ε, το άχυρο, το κάνετε άρρωση και μείνει, τότε μπορεί να δημιουργηθεί περισσότερη λάσπη αργότερα. Αυτό όμως μπορεί να έχει επίπτωση στο υδροφόρο ορίζοντα. Άρα θα δημιουργήσουμε πρόβλημα αν κινηθούμε μόνο στο επίπεδο της οργανικής ύλη. Έπειτα υπάρχουν και άλλα προβλήματα με την οδηγία για τα νητρικά. Μερικά χρόνια είναι τόσο υγρή εισοδιά, ώστε προσπαθώντας καλής να, να θεωρήσει είναι υποχρεωμένος να κάνει έντονη συμπίεση. Αυτό είναι θέμα εποχικό. Τι θέλω να πω. Καλό την Επιτροπή μας αυτό να το κρατήσει έξω από την αρχή της cross compliance. Bene, grazie. Giovanni Lavia ha chiesto la parola. Grazie Presidente. Lama. Λαβία, συγγνώμη. Το πρόβλημα που συζητάμε είναι περίπλοκο. Ευχαριστώ αυτούς που έκαναν τη δουλειά αυτή, ωστόσο υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά κατά περίπτωση ανάλογα με τις συνθήκες του κλίματος και του περιβάλλοντος κατά περιοχή. Δεν είναι δυνατόν να αναλύσουμε αυτό το φαινόμενο παρά μόνο με γενικούς όρους. Μετά θα συζητήσουμε για την κλιματική αλλαγή στο σημείο 4 και την επίπτωση στη γεωργία. Στη Νότια Ευρώπη, Φερρυπίν, τα φαινόμενα που βλέπουμε είναι πολύ διαφορετικά. Χρειάζεται περισσότερο νερό. Το νερό όλο λιγοστεύει και όλο χειροτερεύει. Έχουμε υφάλμηρο νερό πολλές φορές. Οπότε δημιουργείται στήρωση του εδάφους είναι μια κυκλική διαδικασία αυτή. Γι' αυτό πρέπει να το δούμε το θέμα πιο γενικά, πιο καθολικά. Δηλαδή η πολιτική επένδυση να βοηθάει υποδομή η οποία θα επιτρέψει την διατήρηση του νερού, στο χωράφι, προκειμένου να μην χειροτερέψει με τη σειρά του το έδαφος. Δηλαδή, να δούμε όλες τις πτυχές ταυτόχρονα για να έχουμε μια καλή συνολική γεωργική πολιτική που να λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες παραγωγής, όχι μόνο το έδαφος. Ευχαριστούμε τον Τζοβάνι Λαβία, George Lyon και κλείνει αυτός ο κύκλος ομιλητών. Δεν έχει ανοίξει το μικρόφωνο ο That's okay. Thank you. Α, ωραία, ευχαριστώ. Πρόεδρε, έχω να σας πω τα εξή. πρωτα Πρώτα-πρώτα, το θέμα είναι περίπλοκο από πολλές πλευρές. Δύσκολο πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις, γιατί νομίζω ότι σε όλη την Ευρώπη έχουμε χώρες που η καθεμία έχει το δικό της πρόβλημα, τη δική της παραλλαγή του προβλήματος της διάβρωσης του εδάφους ανάλογα με τις πρακτικές, τις διαφορετικές, τις γεωρικές σε κάθε τόπο, και τελικά η λύση ε, πρέπει να αναζητηθεί από τις ε, τοπικές ε, αρχές, τις εθνικές κυβερνήσεις. Εγώ είμαι από την Δυτική Σκότια και άλλα ισχύουν εκεί σε σχέση με ό,τι ισχύει στην Ισπανία. Άλλα ισχύουν Ισπανία και άλλα είναι ο και Σκότια. Επομένω, θα πρέπει η αντιμετώπιση να γίνει σε εθνικό και όχι σε ενωσιακό επίπεδο. Grazie Giorgio. Adesso prima di dare la parola a eh, ancora. Ευχαριστούμε Γιώργο. Λάιον. Πριν δώσουμε το λόγο στον μα και στον Κομισιό, να πω και εγώ δύο λόγια για το σημαντικό αυτό θέμα τη διατήρηση του εδάφου. που κινείται παράλληλα με το θέμα που θα αντιμετωπίσουμε και θα συστήσουμε μετά, δηλαδή την κλιματική αλλαγή. Ο συνάδελφος Στεφάν Λεφόρ θα, μιλήσει, θα μας μιλήσει γι' αυτό. Όλα αυτά έχουν μεγάλη επίπτωση στην ικανότητα νομιμοποίησης της ΚΑΠ στα μάτια όλων των πολιτών. Όποιος θεωρεί ότι η ΚΑΠ πρέπει να συνεχιστεί και μετά το 2013, θέματα όπως το περιβάλλον, η προστασία του εδάφους, η ικανότητα διαχείρισης των φυσικών πόρων, σωστά Όλα αυτά κατά με απαιτούν αυτή την νομιμοποίηση. Και μόνο με την νομιμοποίηση αυτή μπορούμε να ελπίσουμε ότι θα εξακολουθήσουμε να έχουμε υποστήριξη όπως είχαμε μέχρι τώρα εκ μέρους της Ένωσης προς την γεωρική πολιτική. Και τώρα το λόγο στον Γκέι και τον Μονταναρέλα για να απαντήσουν στις ερωτήσεις αν θέλουν. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, μια γρήγορη απάντηση στα συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για τις ε, θετικές παρατηρήσεις σας, ε, για αυτά τα οποία θίξαμε. Υπήρχαν κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις όσον αφορά τον αντίκτυπο της χρήσης ε, ζυζανιοκτώνων κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα γνωστό. Έχουμε δείξει σε πολλές μελέτες ε, το θετικό αποτέλεσμα που έχει αυτή η γεωργία Προστασία του εδάφους και στην βιοπικιλότητα, αλλά οπωσδήποτε δεν υπάρχουν μακροχρόνια εκτεταμένα δεδομένα για την χρήση αυτών των τεχνολογιών σε βάθος χρόνου. Οπότε οπωσδήποτε υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω έρευνα για να ξεκαθαρίσει το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα αυτών των τεχνολογιών. Υπήρχε ένα ερώτημα για το ζήτημα της εντατικής γεωργίας. για το τι μπορεί να γίνει όσον αφορά την διάβρωση. Τώρα όσον αφορά τη μετατροπή χρωτολιβαθικών εκτάσεων σε καλλιεργήσιμη γη βλέπουμε πως υπάρχει αύξηση μόνιμη των δασικών εκτάσεων και της δασοκομείας σε ολόκληρη την Ευρώπη οπότε ίσως υπάρχει κάπου και αντίστροφη τάση για τα υπόλοιπα θα δώσω λόγο συνάδελφο. Κάποιες ερωτήσεις αφορούσαν το επίπεδο πολιτικής αυτό είναι πάντα μια απόφαση που πρέπει να ληφθεί και τονίζει και τις διαφορετικές ευθύνες και επιλογές που υπάρχουν ειδικά στις μελέτες μας ε, στην περιπτωσιολογία βλέπουμε τη σημασία της τοπικής πολιτικής οπότε ίσως σε εθνικό και σε επίπεδο κάτω από το εθνικό να είναι το ιδανικό. Το θέμα είναι ποιος είναι ο ευρωπαϊκός ρόλος, πόσο πρέπει να συντονίζει η Ευρώπη. Όσον αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα, η πολλαπλή συμμόρφωση πράγματι αναφέρθηκε πολλές φορές και προς τις δύο κατευθύνσεις και νομίζω πως ε, αυτό το οποίο έκανε η πολλαπλή συμμόρφωση είναι να το βάλει αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη, να προσανατολιστούμε δηλαδή στο να σκεφτόμαστε τη σημασία του εδάφους Το θέμα δηλαδή πόσο πρέπει να χρησιμοποιηθεί το έδαφος, τι μπορεί να γίνει σε τοπικό επίπεδο, τι σε ευρωπαϊκό. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Και θα συζητηθεί οπωσδήποτε σε αυτό το πλαίσιο, πόσο δηλαδή πρέπει να αναμειχθεί η Ευρώπη, αλλά το σημαντικό είναι ότι τουλάχιστον ετέθη το ζήτημα. Και για τους αγρότες δηλαδή, ότι πρέπει να φροντίζουν το, το χώμα, το έδαφος. Αυτό μπορούμε να πούμε σήμερα. Και τα υπόλοιπα νομίζω ήταν παρατηρήσεις ε, θετικές, ε, μας ικανοποιούν και σας ευχαριστούμε. Bene, cari colleghi, το 4, αν δεν έχετε αντίληψη να το αναβάλουμε και που λέει για την Ευρωπαϊκή και την αλλαγή του είναι ένα θέμα βέβαια πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μα Είναι αυτό το οποίο το είπαμε και προηγουμένω, δηλαδή τι γίνεται με την γεωργική δραστηριότητα, ότι δεν είναι μόνο μέρο του προβλήματο, είναι και μέρο τη λύση. Οπότε, πριν δώσω στον Στέφαν Λεφόλ το λόγο, πρέπει να σα πω ότι έχουμε ζητήσει έγκριση ω Επιτροπή για να κάνουμε έκθεση ιδίας πρωτοβουλία. Βέβαια υπέβαλε ένσταση η Επιτροπή Περιβάλλοντος και είπε ότι θα πρέπει απλώς να συντάξουμε επικουρική γνωμοδότηση Οπότε θα πρέπει να γυρίσουμε συνεπεί σε αυτό που ζητήσαμε και αυτό που κάνουμε σήμερα. Και είπαμε ότι θα πρέπει όσον αφορά την αλλαγή του κλίματο και την γεωργική πολιτική να λάβουμε την έκθεση. Έχει το λόγο ο Στεφάν Λεφόλ. Euh, euh, Πάλι ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αναφέρθηκε ακριβώς η ε, πρωτοβουλία για αυτό το πρόγραμμα και ήταν σωστό αυτό το οποίο ελέγχθη. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται, τι, τι, πώς όλα συμπληρώνονται τα διάφορα επίπεδα αντιμετώπιση σε ενωσιακό, ευρωπαϊκό, κρατικό, τοπικό. Όμως το ερώτημα είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, πώς θα πρέπει να δώσουμε τη λύση ως ε, ασχολούμε με την υγειοργία σε κάθε επίπεδο. Πώς θα απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα. Υπάρχει δεδομένη η αναφέρομαι στο πλανήτη και υπάρχει και ένας μείζον ε, τομέας παραγωγής δραστηριότητα που είναι η ε, παραγωγή ειδών διατροφής. Πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε όσο ασχολούμαι με τη Γεωργία. Πώς μπορεί η Γεωργία να συμμετάσχει, όπως το προηγούμενο ο Ζωζέ. Πώς θα φέρουμε την πτώση της δημοκρασίας του πλανήτη εδώ Τι μπορούμε να κάνουμε τόσο ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις σοβαρές δυσκολίες. Έχουμε παντού πολύ πιο εντό βροχοπτώσει του το οποίο μα οδηγεί σε επιδείνωση τη κατάσταση του εδάφου. Και αυτό γίνεται σε όλο περισσότερα εδάφη, ε, όπου από την άλλη μεριά έχουμε πάρα πολύ σημαντική ξηρασία. Και αυτό αφορά μόνο τι χώρε του Νότου. Αυτό θα σα τονίσω. Και δεν μιλούμε μόνο για Ιταλία και Ανταλουσία. Σύμφωνα με το ΖΙΑΚ, ε, σα λέω έτσι παρεμπιπτόντω, για του συμπατέρε που είναι εδώ, ότι συνολικά η Γαλλία ε, σύντομα πρόκειται να έχει κλίμα καθαρά μεσογειακό. Και επομένω θα πρέπει να αντιληφθούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώ μπορεί να βοηθήσει η Γεωργία σε αυτήν την καταπολέμηση τη ανώδου θερμοκρασία του πλανήτη. Υπάρχουν εδώ πέρα δύο εναλλακτικέ. Η πρώτη είναι το πώ θα αποφύγει η Γεωργία να δημιουργεί αερευλοπτικά που οδηγούν στο δυνατό και αντίστοιχα να προσαρμοστεί η γεωργική παραγωγή. Όλοι σου λένε τα ορυκτά καύσιμα, μιλάμε για πάρα πολύ σήμερα, έχουμε επίσης όλα τα οξύδια του ε, αζότου ε, και έχουμε πάρα πολύ κόσμο που ασχολείται με αυτά ε, και έχουμε επίσης και το μεθάνιο το οποίο παράγουν τα ζώα, εκτινοτροφία. Κάτι το οποίο είναι πολύ πιο βλαπτικό για την ατμόσφαιρα από το διοξίδιο. Άρα έχουμε όλα αυτά τα αέρια τα οποία οδηγούν στην άνοδο της δημοκρασίας. Δεύτερον, πώς η γεωργία, ακριβώς που είναι η γεωργία και που αφορά τους ανθρώπους και τα ζώα, πώς θα μπορέσει να βοηθήσει όσον αφορά ε, τη μείωση του διοξιδίου. Δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να έχουμε λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου. Πρώτα απ' όλα μην έχουμε διαφυγή του αποθεματοποιημένου του διοξιδίου. Και έχουμε εδώ πέρα 70 δις τόνων που είναι αποθηκευμένες στο έδαφο. Οπότε, έτσι θα πρέπει να προχωρήσουμε και στη συνέχεια να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσω της παραγωγής που βοηθάει και στην φωτοσύνθεση. Οπότε να καλύψουν ένα περισσότερο, όλο ένα περισσότερο έδαφος και έτσι να, να παράξουμε όλο ένα και λιγότερο ε, άζωτο ή ε, διοξίδιο. Άλλος παράγοντας εδώ σημαντικός είναι η γεωργία. Εκεί έχουμε ένα τεράστιο χώρο άνθρακα. Άνθρακα που τον χρησιμοποιούμε βέβαια για να ζηταθούμε και έχουμε σήμερα την ε, απογύμνωση της χώρας από τη, τα δάση ε, και αλλού στην Αμαζονία, στην Ιδονησία. Δεν, δεν μπορούν να κάνουν όπως κάνουμε εμείς εδώ πέρα την αναδάσωση. Άρα και έχουν πρόβλημα. επομένω. Ε, εν συνόψη για να ξαναδούμε το θέμα της ανόδου της θερμοκρασίας σε σχέση με το ρόλο της γεωργίας. Ο ρόλος λοιπόν της γεωργίας να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για τη γεωργία και να βοηθήσει να σταθεροποιηθεί το, ο άνθρακα με τις συγκεκριμένε μεθόδους. Και τα δύο στοιχεία αυτά είναι σημαντικά. Υπάρχει ένα τρίτο. Μου το ανάφερε ο πρόσωπο τη Κομισιόν. Η ικανότητα προσαρμογή της γεωργίας στις νέες κλιματολογικές συνθήκες. Ξηρασία, με συγκεκριμένα φυτά που να θίστανται περισσότερο στο υδρικό στρες και αυτό είναι μία παράμετρος που πρέπει να αντιλάβουμε υπόψη μας. Και τελειώνω με ένα πολύ σημαντικό θέμα. Την βιοπικιλότητα. Το λέμε και το λέμε και το λέμε. Να ξέρετε ότι στον 20ο αιώνα 70% της γεωργικής και οικιακής βιοπικιλότητας, δεν μιλάω για τη φυσική, γεωργική βιοπικιλότητα και οικιακή ας το πούμε, βιοπικιλότητα εξαφανίστηκε. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Για να ευνοήσουμε τη βιοπικιλότητα πρέπει να μπορούμε να αναπτύξουμε μοντέλα παραγωγής είτε με σπορά είτε με διάφορες ποικιλίε που θα χρησιμοποιούμε να προωθήσουμε έτσι στην πράξη την βιοπικιλότητα και η βιοπικιλότητα στη γεωργία οδηγεί σε πολλά διαφορετικά γεωργικά προϊόντα που μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε μέσω της αγοράς με προστιθέμενη αξία. Συνοψίζω. Για τη γεωργία και προχώρησε στο πρόγραμμα ΣΟΚΟ πρέπει να έχουμε όλα τα μοντέλα παραγωγής που να επιτρέπουν να μειωθεί η κατανάλωση της ε, ορυκτής ενέργειας, των αερίων θερμοκηπίου, που, μοντέλα που θα επιτρέψει τη γεωργία να φυξάρει να σταθεροποιεί τον άνθρακα, άρα να μειώνονται τα αέρια θερμοκηπίου και τρίτον η γεωργία να μπορεί να βοηθάει ταυτόχρονα και τη βιοπικιλότητα και όπως είπε ο πρόεδρος μας πριν που είναι πολύ σημαντικό να είναι μια κοινωνική παράμετρος της απάντησης που θα φέρουμε στο ερώτημα της κλιματικής αλλαγής. Αύριο αυτό θα δικαιολογεί το ότι θα μπορούμε να έχουμε ακόμα μια κοινή γεωργική πολιτική. Σας ευχαριστώ. Bene, grazie Uh... Πρόεδρος, σε ευχαριστούμε Στεφάν. Και αρχίζει η συζήτηση για το σημαντικό αυτό θέμα. Κύριε Μπότσον πρώτη. Μπότσον, madame. Tack, herr ordförande, och tack, föredragande. Er ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή. Νομίζω πως ασχολούμαστε τώρα με τα δύο σοβαρότερα ζητήματα ε, για το παρόν και το μέλλον της ε, Γεωργίας. Και είναι δική μας ευθύνη το ότι πρέπει να ασχοληθούμε με το κλίμα, με τη γεωργία, με το πώς θα κινηθεί τώρα η διαδικασία έτσι ώστε και ο Ευρωπαίος πολίτης να αντιληφθεί πως η γεωργία δεν είναι ο μεγάλος κακός εδώ πέρα όσον αφορά την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Αντιθέτως είναι ο σημαντικότερος παράγοντας της λύσης των τεράστιων αυτών ε, προβλημάτων. Τα προβλήματα της ε, κλιματικής αλλαγής ανεξαρτήτως του ποια είναι η αιτία θα μας οδηγήσουν στο να έχουμε πιο ξηρά μέρη εκεί που είναι ήδη ξηρά, πιο υγρά εκεί που είναι ήδη υγρά. Γνωρίζουμε πως ε, θα έχουμε αρρώστιες, ε, γιατί θα υπάρχουν οι φορείς αυτών των ε, ασθενειών, ειδικά σε εμά το βορρά, είναι πιο ζεστοί οι χειμώνες. Γνωρίζουμε πως ένα τμήμα του προβλήματος είναι το μεθάνιο και το άζωτο. Κοίταξα εγώ την έρευνα και μπορώ να θυμηθώ εγώ κανείς δεν μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα είτε μιλάμε για κοπριά είτε για λιπάσματα πόσο είναι αυτό το άζωτο που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Οπότε δεν υπάρχει αρκετή έρευνα. Το άζωτο είναι 230 φορές πιο επικίνδυνο από το διοξίδιο του άνθρακα. Ναι, διαφύλαξη του εδάφους, ναι, προστασία του εδάφους. Εάν μπορούσαμε να αυξήσουμε τη φωτοσύνθεση και τη σοδιά ταυτόχρονα, εάν μπορούμε να δεσμεύσουμε περισσότερο του άνθρακα στο έδαφος, να αποθηκεύσουμε, τότε θα μπορέσουμε να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Και υπάρχει και το πρόβλημα των εντομοκτώνων, των ζυζανιοκτώνων, καθώς η έρευνα σήμερα βρίσκεται στα χέρια των τεράστιων ε, χημικών εταιριών. Πού είναι η ανεξάρτητη έρευνα, τη χρειαζόμαστε. Τη χρειαζόμαστε απεγνωσμένα στη γεωργία. Χρειαζόμαστε ζανιοκτώνα που δεν θα είναι δηλητηριώδη, μάλλον θα είναι δηλητηριώδη εκεί όπου πρέπει να είναι. Και μετά όχι. Και υπάρχει και μια τρίτη πτυχή δηλαδή η παραγωγή ενέργειας. Έχουμε τεχνολογία, επίκαιρη τεχνολογία και με την ε, βοήθεια της τεχνολογίας θα πρέπει να είναι αυτόνομη η γεωργία όσον αφορά ε, τη γεωργία. Δεν χρειάζεται κανείς να αγοράζει δίζελ αν έχει τόσο πολύ βιομάζα. Έχουμε την τεχνολογία, γνωρίζουμε την τεχνολογία, ξέρουμε πώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ζήτημα μόνο πολιτικής βούλησης, οπότε δεν είναι πλέον θέμα Έρευνα Γνωρίζουμε πώς έχουν τα πράγματα και εάν μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη φωτοσύνθεση, εάν μπορούμε να δεσμεύσουμε περισσότερες τέτοιες ουσίε από τον αέρα, έχουμε το υλικό με το οποίο μπορεί να παραχθεί ενέργεια και υπομορφή καυσίμων, αλλά και ρεύμα μπορούμε να και σε ρεύμα μπορούν να μετατραπούν αυτές οι, οι πηγές ηλεκτρικό οπότε νομίζω πως ε, ο ρόλος της γεωργίας θα πρέπει να εδραιωθεί πάλι ως ε, το κύριο τμήμα της λύσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την ενδιαφέρουσα έκθεσή του και συμφωνώ πράγματι είναι σημαντική η κλιματική αλλαγή για τη γεωργία και το γεγονός ότι η γεωργία θεωρείται μέρος του προβλήματος είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που θα πρέπει να δώσουμε στον κλάδο σύντομα αλλά ταυτόχρονα η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι πως η γεωργία μπορεί να αποτελέσει μέρο τη λύση. Και από αυτή την έννοια σημαίνει αυτό πολλές ευκαιρίες για τη γεωργία. Τώρα κοιτώντα το μέλλον δεν θα είναι εύκολο αυτό γιατί θα συνδεθεί με την αυξανόμενη ζήτηση για να ταΐσουμε τον παγκόσμιο πληθυσμό που αυξάνεται συνεχώς. Οπότε πώς θα συνδυαστεί αυτό με τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και του της αύξησης του πληθυσμού. Και βέβαια το ζήτημα είναι τι ρόλο μπορεί να παίξει το, το κράτος. Και όπως και με το προηγούμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, όσον αφορά την νομοθεσία, οπωσδήποτε η νομοθεσία θα πρέπει να θεωρείται η τελευταία λύση και να έχουμε ελαφρές επεμβάσεις και είμαι πεπισμένος πως το κλειδί εδώ πέρα είναι η έρευνα και η ανάπτυξη και θα ήθελα να το συμπεριλάβει ο εισηγητής. Έχει υπάρξει τραγική μείωση των πόρων που αφιερώνονται σε έρευνα των ζητημάτων αυτών και για το προηγούμενο ζήτημα της ημερήσιας διατάξης και για αυτό και πρέπει να ζητήσουμε περισσότερη κρατική στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης όλου του κλάδου. Ευχαριστώ, George Lyon. Έχει ε, ζητήσει τον λόγο. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα. Συμφωνώ και εγώ με αυτά που είπε στην Άρφο Σάσκοροφ. Οι κλιματολογικέ αλλαγέ, όπως λέει και ο εισηγητή, είναι μια από τι πιο σημαντικέ αλλαγέ και η Γεωργία καλείται να παίξει ρόλο στο μέτωπο αυτό. Είναι κομμάτι της λύση. Η παραγωγή του μεθανίου μέσω των ζώων είναι μια σοβαρή πρόκληση. Πρέπει να βρούμε λύση. Και ξαναγυρίζουμε σε αυτό που είπε ο Ρίτσαρντ. Πρέπει να γίνει έρευνα προκειμένου να βρεθούν μέτρα που να μετριάζουν την κατάσταση. Η Νέα Ζηλανδία έχει προχωρήσει πολύ στο θέμα αυτό. Έχει υπάρχει μια μείωση εκεί στα μυρικαστικά, γύρω στο 10% στις εκπομπές, αλλά χρειάζονται επενδύσεις, χρειάζονται επενδύσεις και στον υπόλοιπο κόσμο, προκειμένου να βρεθούν λύσεις στο πρόβλημα. Είναι πολύ δύσκολο το θέμα των εκπομπών μεθανίου εκ μέρους των ζώων. Έπειτα πρέπει να μειωθεί η ενέργεια που χρησιμοποιεί η γεωργία. Το 1% της παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας χρησιμοποιείται στη γεωργία με παραγωγή λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, καύσιμα. Πρέπει να αναπτυχθούν καλλιέργειες και φυτά που να μπορούν να καλλιεργούνται με λιγότερη ενέργεια. Αυτό σημαίνει έρευνα και κρατική έρευνα για νέα φυτά που να χρειάζονται λιγότερο άζωτο, λιγότερα φυτοφάρμακα, λιγότερη ενέργεια. Δυστυχώς αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή οι εμπορικές εταιρείες ασχολούνται μόνο με το θέμα, οι κυβερνήσεις όχι. Χρειάζεται λοιπόν έρευνα και ανάπτυξη εκ μέρους του δημοσίου, προκειμένου να δοθούν μέτρα μετριασμού του προβλήματος, όσον αφορά τα φυτά και όσον αφορά τα ζώα. Ελπίζω στην έκθεση ο συνάδελφος να τονίσει αυτή την ανάγκη για έρευνα και ανάπτυξη προκειμένου να μειωθεί η επίπτωση του άνθρακα, του carbon input. Μάρτιν Όσλιμ. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Πράγματι αναφέρθηκαν σημαντικά ζητήματα και τα υποστηρίζω πάρα πολύ. Η γεωργία αφενός είναι και θύμα αλλά και προκαλεί ταυτόχρονα μεταξύ άλλων βεβαίω στην κλιματική αλλαγή. Αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση ενέργειας όσον αφορά τη χρήση καυσίμων αλλά και δευτερογενώ ε, με την χρήση καυσίμων για συνθετικό άζωτο παραδείγματο χάρη οπότε πρέπει να τα λαμβάνουμε όλα αυτά υπόψη αν είναι να σκεφτούμε πώς και η γεωργία θα συνεισφέρει στη μείωση της κλιματικής αλλαγής. Εγώ θεωρώ πως ε, πρέπει να εμπλακεί και η Γεωργία οπωσδήποτε τα επόμενα χρόνια να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα μειώσει τους ε, στόχους όσον αφορά το, το κλίμα για να συνεισφέρουμε και εμείς στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Ε, δεύτερον, το οποίο πρέπει να συζητήσουμε πολύ σοβαρά και οπωσδήποτε δεν το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, είναι το θέμα του μεθανίου. και ηλεκτρικό αέριο γιατί υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ε, τέτοιες εκπομπές ε, από τη Γεωργία, κάτι το οποίο οφείλεται και στην ε, μεγάλη χρήση λιπασμάτων. Και οπωσδήποτε πρέπει εδώ πέρα να παίξει τον ρόλο της η Γεωργία. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε ξανά μια περιφερειακή έτσι κυκλοφορία, ένα περιφερειακό κύκλο όσον αφορά την χρήση της ενέργειας. Δεν είναι ανάγκη να μεταφέρονται τα προϊόντα από την μία άκρη της Ευρώπης στην άλλη για να κατανοηθούν, αν υπάρχει μια τοπική δυνατότητα. Πρέπει να δούμε λοιπόν και το ζήτημα της μεταφοράς των προϊόντων και αυτό θα πρέπει να εμποδιστεί στο μέλλον. Και επειδή κάποιος είπε πως, επειδή ο ΙΕ είπε πως εμείς δεν έχουμε προβλήματα στην Ευρώπη, τα προβλήματα τα έχουν στην Νότια Αμερική, το έχουμε προκαλέσει εμείς αυτό το πρόβλημα, γιατί μεγάλο τμήμα των ζωοτροφών προέρχονται από την Λατινική Αμερική. Εάν δούμε τι, τι γίνεται και πού καταναλώνονται αυτά, είναι άρα πρόβλημα και της δικής μας ε, γεωργίας. Οπότε αν δεν ήταν αυτή η παραγωγή στην Νότια Αμερική θα γινόταν εδώ πέρα. Οπότε πρέπει να δούμε μήπως θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε π.χ. παραγωγές ε, φυτικών ε, λευκομάτων ε, και στην Ευρώπη για να χρησιμοποιηθούν στις ζωοτροφές. Οπότε σε ένα πράγμα συμφωνούμε Χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα που θα βασίζεται σε πραγματικά επιστημονικά στοιχεία για το μέλλον της ε, γεωργίας όσον αφορά την συνεισφορά μας στην μείωση της κλιματικής ε, αλλαγής. Αυτό πρέπει να ενισχύσουμε. Και εγώ θα συμφωνήσω με τον Μάρτιν και σας καθισγάζω λέγοντά σας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη την επιφάνεια η οποία χρησιμοποιούνται αυτά τα 50 εκατομμύρια τόνων που εισάγονται στην Ευρώπη που αντιστοιχούν σε 20 εκατομμύρια εκτάρια. Δηλαδή ένα πρόβλημα του κλιματικού προβλήματος σε σχέση με τη γεωργία αυτό εξωτερικεύεται με τις άλλες, προς τις άλλες χώρες. Άρα έτσι θα προχωρήσει η προβληματική μας για να λάβουμε υπόψη το πώς είναι δομημένη η κτηνοτροφία και τι είδους ζωικές πρωτεΐνες εισάγουμε. Άρα, το τι γίνεται με τις πρωτεΐνες στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντική κουβέντα που μας οδηγεί στο να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε κάποια κυκλική εναλλαγή στις καλλιέργειες άλλο σημαντικό το οποίο πολλοί ανέφεραν είναι το μεθάνιο. Και εδώ υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες να το ξαναχρησιμοποιήσουμε στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις ε, τοπικές κοινότητες. Ε, γίνεται αυτό όπως στην Γερμανία, στην Αυστρία επίσης και σε πολλές χώρες. Όμως ε, ακόμα δεν γίνει τίποτα, βρίσκονται πίσω αυτές οι χώρες, υπάρχουν όμως δυνατότητες και αυτό μπορεί να γίνει μέσα στη γεωργική εκμετάλλευση, την οικογενειακή. Εξορθολογιστικά, εξορθολογισμένα και κάτι άλλο που μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό, το κλίμα όπως ε, ανεφέρθη, ε, επηρεάζεται από τις γεωργικές πολιτικές με διαφορετικές σε κάθε τρόπο και επίσης είναι και ένα θέμα του τι σπόροι χρησιμοποιούνται. Δεν είναι απλώς θέμα στα τεχνολογική Είναι και το θέμα του να μπορεί να ληφθεί υπόψη από μια συμμετοχική έρευνα το πώς εξελίσσονται, πώς μπορούν να εξελιχθούν οι σπόροι που χρησιμοποιεί η εκμετάλλευση. Άρα να γίνει ανάπτυξη σε αυτό το σημείο. Οι σπόροι που παρουσιάζονται μέσα στην ε, ε, επιχείρηση, την εκμετάλλευση και αυτό αλλάζει χρόνο με χρόνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήξερες τον κανόνα. Από το 98 έχουμε βελτίωση. Και ας μην το δέχεται ο κόσμος. το Φεβρουάριο είχα πάει στην Ινδία. Το Φεβρουάριο του 2008. Κοιτάξτε, άνθρωποι 60 χρονών έλεγαν πως είναι ο πιο κρύος χειμώνας που είχαν δει ποτέ. Πέρσι, 08-09. Έξι συνεχόμενοι μήνες χιόνι. στο δικό μου αγρόκτημα, στην Ανατολική Αγγλία. Οπότε αν ε, έχουμε πρόβλημα παγκόσμια θέρμανσης, εγώ δεν το βλέπω. Κοιτάξτε, τα αέρια του θερμοκηπίου, θα δούμε ποιο είναι το μεγαλύτερο. Είναι οι υδρατμοί. 70%. Δεν μπορούμε να κάνουμε όμως ε, τίποτα. Τι θα κάνουμε για του υδρατμούς. Τίποτα γιατί του χρειαζόμαστε. Οπότε καταλήγουμε στο διοξείδιο του άνθρακα. Πόσοι γνωρίζουν πω είναι 0,038 τη ατμόσφαιρας. Αυτό είναι όλο. Είναι 10 φορέ περισσότερο. Ε, ήταν 10 φορέ περισσότερο στο παρελθόν και όταν ήταν περισσότερο ήταν πιο κρυο ο καιρό. Εγώ το χρειάζομαι. Είμαι αγρότη για να αναπτυχθούν τα προϊόντα μου. Οπότε μην το ξεχνάμε. Μεθάνιο. Πόσο υπάρχει στην ατμόσφαιρα. 0,0000002%. Δεν είναι και πολύ έτσι. Και αν σκεφτούμε πως το, μεγαλύτερο από αυτό, παράγει, το περισσότερο από αυτό παράγεται από οργανισμούς των πυθμένα. Και μην καταστρέψουμε τώρα και τα μυρικαστικά, είναι μέρος της ζωής με, το, με τις αχλαμάρες αυτές. Συμφωνώ τώρα για το άζωτο. Ναι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λιγότερο άζωτο εάν χρησιμοποιήσουμε βιοτεχνολογία, γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Αλλά οι περισσότερο πέρα το θεωρούν κάτω διαβολικό, κακό κτλ. Οπότε ούτε αυτό μπορούμε να κάνουμε. Μια κουβέντα για τη σόγια και την πρωτεΐνη. Πράγματι το εισάγουμε, συμφωνούμε, εισάγουμε πάρα πολύ σόγια θα μπορούσαμε βεβαίω να παράγουμε πολύ περισσότερη πρωτεΐνη δική μα στην Ευρώπη αν χρησιμοποιήσουμε βιοτεχνολογία. Είτε μπορούμε να τα προσαρμόσουμε τη σόγια δηλαδή για να αναπτύσσεται σε ψυχρότερα κλίματα ή τα δικά μας τα ψυχανθεί για να έχουμε σοδιά κάθε δύο χρόνια αντί για κάθε έξι χρόνια. Αυτά και ε, αντιλαμβάνω πως είναι εξαίρεση στον κανόνα. Ευχαριστώ, Γκλατφέλτερ. Ναι, ευχαριστώ. Εγώ θέλω να σας επισύρω την προσοχή στο εξής. Θεωρούμε ότι αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, οπότε και θα πρέπει να τονίσουμε το πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έχοντας τέτοια πολιτική εξοικονομής ενέργειας σε όλους τους τομείς. Στην Ουγγαρία η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έτσι δεν εκμεταλλευτήκαμε τους ευρωπαϊκούς πόρους ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ανανεώσιμους ε, ενεργειακούς πόρους. και προσπαθούμε και στον τομέα της παραγωγής τροφίμων αλλά και στη γεωργία να έχουμε τέτοια φιλική στον περιβάλλον πολιτική. Όμως τι θα γίνει μετά το 2013 γιατί θα είναι πάρα πολύ σημαντικό με το προπολογισμό οι ανανεώσιμες σπίσεις ενέργειας, η εξονόμηση ενέργειας και στην παραγωγή τροφίμων αλλά και στη γεωργία. Όμως πρέπει να προσέξουμε και κάτι άλλο. Υπάρχει κάποια αντίφαση πάρα πολύ συχνά. Θεσπίζονται κάποιοι κανόνες και με αυτούς τους νέους κανόνες η γεωργία καταναλώνει περισσότερη ενέργεια. Φερρυπίν, θέλω να σας παραπέμψω στην νομοθεσία για την καλομεταχείριση των ζώων. Οι και οι καλομεταχείριση των ζώων οδηγούν σε περισσότερη κατανάλωση ενέργεια. Επομένω, στο μέλλον δεν θα πρέπει να πέφτουμε σε αυτό το λάθο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την κλιματική αλλαγή εγώ είμαι πάντα πολύ προσεκτικός γιατί αν δούμε τα δύο τελευταία 2.000 χρόνια και στο παρελθόν είχαμε σοβαρές κλιματικές αλλαγές. Απλά δεν υπήρχε τηλεόραση. Αποδεδειγμένο... Αποδεδειγμένα υψηλότερη στάθμη των νερών στην Ευρώπη ήταν το 1342 τι έφταιγε τότε το διοξείδιο του άνθρακα. Οπότε υπάρχουν πάντα αλλαγές ε, στο, στο κλίμα. Σας είπα ποια ήταν η υψηλότερη σταθμή του νερού στην Ευρώπη και πλημμύρες ε, υπάρχουν πάντα όταν βρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Απλά είναι τα παραγμάτα και αν δούμε και τη στάθμη των ε, ποταμών στη Βαβαρία και την Αυστρία ε, έχουν φτάσει σε πολλού αιώνες στο παρελθόν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα χωρίς να θέλω να πω πως δεν υπάρχει κανένα κίνδυνος. Απλά πρέπει να μην ξεχνάμε πως υπάρχουν εδώ πέρα και νέα οικονομικά συμφέροντα που κρύβονται από πίσω και βεβαίως πράγματι θα πρέπει να έχουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερες γεές στην διάθεσή μας και οπωσδήποτε η γεωργία δεν είναι εδώ πέρα αυτή η οποία καταστρέφει το κλίμα, καλά το είπε η συνάλφος, εμείς μπορούμε να συνεισφέρουμε στη μείωση εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα όπως σας είπα εγώ για το σπίτι μου χρησιμοποιώ κάθε χρόνο 7.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ε, και το έχω αντικαθαστήσει πλέον με απορρίμματα ξύλου και δεν χρησιμοποιώ πλέον αυτό το πετρέλαιο θέρμανσης. Οπότε μπορούμε με έρευνα και με επιστήμη να αντικαταστήσουμε πάρα πολλά πράγματα και θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να ερευνήσει

να εκμεταλλευτούμε την ε, βιομάζα ειδικά στα κτίριο. Να σκεφτούμε και όταν είναι π.χ. ξύλινα τα παράθυρα και... και τα δοκάρια του σπιτιού και οτιδήποτε, ε, όπως το δικό μου το σπίτι που είναι 400 ετών, 400 χρόνια δεσμεύουν εκεί πέρα διοξίδιο του άνθρακα κατασταθούν όλες αυτές οι τεχνικές, οι συνθετικές ουσίες από ξύλινα κουφώματα παραδείγματο χάρη. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Χρειάζεται όμως οπωσδήποτε έρευνα και μπορούμε να έχουμε και πρακτικές λύσεις ε, για τη γεωργία συμπεριλαμβανωμένη στις δασοκομείς για να συνεισφέρουμε στο κλίμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλμπερτ, κυρία Ντότσου. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φαίνεται πως υπάρχει μια σοβαρή συζήτηση για το εάν υπάρχει πραγματικά θέρμανση του κλίματος ή μια κυκλική αλλαγή του κλίματος. Αλλά όποιες και αν είναι οι απόψεις σας επ' αυτού, Υπάρχουν κάποια πράγματα που θα πρέπει να θυμόμαστε ε, σε σχέση με τους αγρότες. Στη Βόρεια Ιρλανδία, από όπου κατάγομαι εγώ, οι περισσότεροι αγρότες είναι μικροί, οι εκμεταλλεύσεις είναι οικογενειακές και θεωρούν πως διαφυλάσσουν το περιβάλλον. Θέλουν να παραδώσουν καλό περιβάλλον και στις επόμενες γενιές που είναι τα παιδιά τους. Καθώς η εκμετάλλευση μένει στην ίδια οικογένεια για γενιές και είναι προς το συμφέρον τους να παραδώσουν κάτι πολύτιμο και σωστό και αηφόρο για το μέλλον. θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ασχοληθεί με δύο ζητήματα. Το ένα είναι πως πρέπει να το δούμε σε εθνικό επίπεδο αυτό το θέμα για να μπορέσουμε να εξετάσουμε τους διάφορους τρόπους και τα συστήματα παραγωγής που ισχύουν ε, όχι μόνο σε διαφορετικά σημεία της Ευρώπη, αλλά και σε διαφορετικά σημεία της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδία. Π.χ. στη Βόρεια Ιρλανδία ε, ο τομέας ε, της γαλακτοπαραγωγή βασίζεται κυρίως στο σχορτόλιβαδικές εκτάσεις που θα μας έδινε ίσως εάν το μετρούσαμε περισσότερο υψηλό ποσοστό μεθανίου σε σχέση με άλλες πιο εντατικές όμως ε, μεθόδους. Οπότε όποιο και να είναι το αποτέλεσμα των συζητήσεων πρέπει να θυμόμαστε πως δεν θα πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για περαιτέρω γραφειοκρατία και ρυθμίσεις. Και πως οι μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές για τους αγρότες σε αυτό το κλίμα της οικονομικής ε, δυσπραγίας είναι πέρα από τις δυνατότητες των αγροτών. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε πρακτικές προτάσεις και να μην οδηγηθούμε πάλι σε νέες οδηγίες. Διακριτικά όσον αφορά τις ρυθμίσεις ε, στην ε, Γεωργία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τον λόγο έχει ζητήσει ο κύριος E, to niezwykle ważny dokument e, i oczywiście można... Οι γεωργοί το καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά αυτές τις συζητήσεις. Το πρόβλημα είναι πώς να βοηθήσουμε τους γεωργούς για να καταλάβουν και να προσαρμοστούν στις αλλαγές αυτές είτε όσον αφορά την παραγωγή της επιμέρους γεωργικής εκμετάλλευσης, διότι πολλοί γεωργοί σήμερα έχουν προβλήματα εφοδιασμού με νερό, διαχείριση λοιπόν των, των υδάτων, των αποβλήτων, των εκμεταλλεύσεων. Όλα αυτά βέβαια τα αναφέρει η έκθεση. Επίσης πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Γεωργία είναι leader όσον αφορά την καταπολέμηση των κλιματολογικών αλλαγών. Όταν μιλάμε λοιπόν για κλιματολογικές αλλαγές, πρέπει να με αυτό το πνεύμα να προγραμματίσουμε τη μελλοντική ΚΑΠ. Βέβαια χρειάζεται πολλή έρευνα, πολλή ανάλυση, Όσον αφορά όμως την τρέχουσα κατάσταση πρέπει να αξιοποιήσουμε όσα στοιχεία έχουμε μέχρι τώρα από την έρευνα. Έπειτα, πώς χρησιμοποιούμε τα κονδύλια της Ένωσης για την ανάπτυξη της υπαίθρου για να αυξηθεί η καλλιεργούμενη περιοχή των δασών στην Ένωση. Τα κονδύλια αυτά βοήθησαν τους γεωργούς, επέτρεψαν την καταπολέμηση των κλιματολογικών αλλαγών μέχρι τώρα Έπειτα η ανάλυση όλων αυτών των εγγράφων και κειμένων, όλων αυτών των ερευνών, πρέπει να επηρεάσουν θετικά τον μελλοντικό προγραμματισμό της ΚΑΠ. Αυτό είναι δουλειά μας, της Επιτροπής Γεωργίας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, ξέρετε, πως, όπως ξέρετε στη χώρα μου 70% της έκτασης είναι κάτω από το ύψος της ε, θάλασσας και όταν ζει βεβαίως κάποιος 6 ε, μέτρα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας δεν μπορεί να εμπλακεί σε ακαδημαϊκή συζήτηση για το εάν υπάρχει τέτοια αλλαγή του κλίματος. Πρέπει να έχουμε μια επιτυχία στην Κοπενχάγη όσον αφορά τη Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή. Αυτό το οποίο με ενοχλεί είναι πως ε, και στη δική μου τη χώρα φαίνεται πως η γεωργία είναι ο μόνος ένοχος να μιλάμε για την κλιματική αλλαγή και μας λένε κάθε εβδομάδα να γίνουμε όλοι χορτοφάγοι για να σώσουμε το κλίμα, ενώ πετάμε κάθε εβδομάδα 20 έως 30% ε, του φαγητού και εγώ θα ανισχούσα πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή που γίνεται στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για το λεγόμενο αποτύπωμα άνθρακα τα αυτοκόλλητα που μπαίνουν στα τρόφιμα και μπαίνουν σε κάποιο σούπερ μάρκετ π.χ. το Τέσκο έχει τον δικό του ορισμό και βάζει δικές του ενδείξεις οπότε πλέον δεν αξίζει τίποτα αυτή η σήμανση. Οπότε το θέμα είναι ακριβώς ο ορισμός ε, γιατί εντάξει το πώς θα γίνει αυτός ο ορισμός, το ποιος θα δίνει αυτό το αυτοκόλλητο, το ποιος θα αξιολογεί το αποτύπωμα αυτό διοξείδιο του άνθρακα είναι σημαντικό, αλλά να μην έχουμε πάρα πολλέ και άρα τελικά χωρί κανένα νόημα πρωτοβουλία. Οπότε επίση θα πρέπει να σκεφτούμε και πρωτοβουλίε για το πώ θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί και να αποθηκευτεί υπόγεια το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτή την καινοτομία πρέπει να τονίσουμε και για τη μελλοντική πολιτική και αυτή τη στιγμή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το διοξείδιο του άνθρακα για να κερδίσουμε και θερμότητα και ενέργεια, αλλά λένε μεγάλε ευκαιρίε, είναι πολύ μικρές αυτές οι ποσότητε, δεν μα ενδιαφέρουν, οπότε σταματάει η έρευνα σε αυτόν τον τομέα. Αλλά αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι αυτό το οποίο μας απασχόλησε και πριν, δηλαδή η βιοπικιλότητα, γιατί αυτό ε, η κλιματική αλλαγή θα έχει επιπτώσει και στη βιοπικιλότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το είπε ίδια πριν από λίγου μήνε σε μια εκθεσή τη. Τα μέσα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη για να εργαστούμε για τη βιοπικιλότητα είναι πάρα πολύ στατικά. Η βιοπικιλότητα, η σχετική νομοθεσία όπω ορίζεται στην οδηγία για τα πτηνά και για τους ε, βιοτόπους είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Δηλαδή λέμε εδώ πέρα υπάρχει το χύψη φυτό ή ζώο, γύρω γύρω κάνουμε ένα κύκλο και έτσι θα το προστατεύσουμε. αλλά βλέπετε τι γίνεται και τα ζώα και στα Πυρηναία και στην Νότια Σουηδία. Επηρεάζονται ήδη άμεσα τα ζώα από την κλιματική αλλαγή, αλλάζουν τους βιοτόπους τους. Οπότε θα πρέπει και η νομοθεσία μας να δούμε τι γίνεται, γιατί δεν είναι εξοπλισμένη να απαντήσει σε αυτά τα φαινόμενα. Δεν ξέρω εάν ακόμα ενδείκνυται αυτή η στατική προσέγγιση την οποία έχουμε. Θα πρέπει να πάμε σε μια πιο δυναμική αντιμετώπιση. Αυτά για το μακροπρόθεσμα και λέω πως ε, θα ήθελα και εμείς να λάβουμε μέρος σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Θα τελειώσουμε τη συζήτηση με τον ε, Αντιπρόεδρο κ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι για την ε, συζήτηση αυτή, αλλά πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα γιατί πράγμα μιλάμε. Πριν από πέντε χρόνια, όταν ξεκίνησε τη θητεία του το προηγούμενο κοινοβούλιο, μιλούσαμε συνεχώς για global warming, θέρμανση του πλανήτη. Τώρα ξαφνικά μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Στο παρελθόν μιλούσαμε για θέρμανση, υπενθυμίζω. Και σε λίγα χρόνια βλέπετε θα μιλάμε ε, για κάτι τελείως διαφορετικό, για την ψύχρανση του πλανήτη. Δεν ε, είμαι ειδικό, δεν θα ε, αντιδαχθώ εγώ στους ειδικού που λένε ότι αλλάζει πράγματι το κλίμα και ότι μπορεί να το επηρεάσει ο άνθρωπος, αλλά ακούω και άλλες φωνές που λένε πως ε, όλα αυτά είναι τελείως ε, αστήρικτα. Το ανέφερε και ο συνάδελφος, πάντα υπήρχαν κλιματικές αλλαγές, πάντα άλλαζε και αλλάζει το κλίμα και ο άνθρωπος δεν είχε καμία επίδραση στο παρελθόν. Και νομίζω και σήμερα ε, εξίσου λίγη επίδραση έχει. Οπότε πρέπει να το πούμε αυτό ξεκάθαρα σε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή έχουμε ελάχιστη γνώση σε αυτόν τον τομέα, γιατί έχουν αίσθηση πως εδώ πέρα μιλάμε για κάτι το οποίο δεν είναι απολύτω σίγουρο. Εγώ εκπροσωπώ μια χώρα η οποία θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις ε, από αυτά τα νομοθετήματα στο πλαίσιο της ε, κλιματικής αλλαγής. Η βιομηχανία μας όπως ξέρετε πρέπει να μειώσει τι εκπομπέ τη κατά 30% σε σχέση... Τι μείωσε ήδη από το 1990 και πρέπει τώρα να τι μειώσει ακόμα περισσότερο. Και τώρα μιλάμε και για τη γεωργία από που πρέπει να βοηθήσει η γεωργία στην κλιματική αλλαγή. Είναι δύσκολο να αποδεχτούμε κάτι τέτοιο. Κύριε Πρόεδρε, θυμάμαι εγώ ακόμα πως ε, δεν είχαμε εμείς ε, π.χ. στο χωριό μου καθόλου εκπομπές ε, αλλά δεν είχαμε και καθόλου τρακτέρ. Δεν ξέρω αν θέλουμε να επιστρέψουμε σε μια τέτοια εποχή. Πριν δώσω το λόγο στην Κομισιόν και αφού είχαμε μια ευρεία συζήτηση με πολλές διαφορετικές απόψεις και ευαισθησίες όπως τις ακούσαμε να εκφράζονται οι κλιματολογικές αλλαγές είναι ένα θέμα που αφορά την Επιτροπή μας. Αφορά το μέλλον της γεωργίας. Και όπως κάποιος είπε, είναι τμήμα του προβλήματος, αλλά είναι και τμήμα της λύσης. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε έναν έξυπνο τρόπο να χειριστούμε το δύσκολο αυτό θέμα και ο Στάφος Στεφάν Λεφόρ θα κάνει την έκθεση και ελπίζω τελικά όλοι να βρεθούμε στο ίδιο μήκος κύματος το λόγο στους εκπροσώπους της Κομισιόν. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα σα πω ότι με μεγάλη μα χαρά ακούμε την πρόταση για τη σύνταξη εκθέσεως ιδίας πρωτοβουλίας. Είμαστε σίγουροι θα βοηθήσει για το δικό μας έργο σε σχέση με την μεταρρύθμιση της ε, κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής για το 2013 και μετά. Έχουμε τις ε, προπαρασκευαστικές ε, σκέψεις, για τις γραμμές, έχουμε σχετικά δύο έγγραφα εργασία που φέτος παρουσιάσαμε και όσον αφορά την προσαρμογή δηλαδή της γεωργίας στην του κλίματος και από την άλλη μεριά τις δυνατότητες που υπάρχουν ώστε να μειωθεί αυτό το φαινόμενο σε σχέση με τη γεωργία και τα βασικά σημεία ήδη έχουν τονιστεί. Αυτά τα εξετάζουμε και εμείς σε αυτά τα δύο εγγραφά μας. Πρώτα-πρώτα έχουμε κάποιες ε, αναπόφευτες αλλαγές στο κλίμα. Αυτά έχουν παρατηρηθεί, αυτά εξελίσσονται σαν φαινόμενα και βέβαια πρόκειται για κάποια πλήγματα που δέθηκε η Γεωργία. είναι τάση πια καθιερωμένη, τον έχουμε κάποια κρύα φαινόμενα. Οπότε έχουμε έτσι ζημία ο πλευράς Γεωργών. Και η επιστήμη βεβαιώνει ότι αυτή η τάση βαίνει αυξανόμενη. Εμεί παρουσιάσαμε ένα πλαίσιο δράση, εκείνη την λευκή βίβλο για την προσαρμογή στο κλίμα την σου χαρακτήρα, αυτό το έγγραφο και πάντως τονίσαμε τις ε, πτυχές που αφορούν τη Γεωργία. Η Γεωργία φυσικά δεν χρειάζεται εμάς να κάτσουμε να τους πούμε πώς θα προσαρμοστούν στα καιρικά αυτά φαινόμενα. Γιατί κάθε μέρα τα αντιμετωπίζουν. Όμως, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον πρόθεσμα μπορούμε να προβλέψουμε κάποιες αλλαγές που θα γίνουν, αλλά ίσως δεν ξεπερνούν τους Γιώργους. Άρα, τουλάχιστον για ανταλλαγή εμπειρίας και για έρευνα, μπορεί η Ευρώπη να βοηθήσει. Και έτσι, περιφερειακές και τοπικές συνθήκες, υπάρχει περίπτωση να βοηθήσει καθόλου τον τρόπο η Ευρώπη. Έχουμε άλλωστε και τις εκπομπές, των αερίων του θερμοκηπίου και όπως προαναφέρθηκε δεν είναι ο βασικός ενοχός η Γεωργία γιατί από το 1990 μειώνονται οι εκπομπές στην Ευρώπη και τώρα φτάσανε σε επίπεδο πολύ χαμηλότερο σε σχέση με ενεργειακό τομέα, με βιομηχανία, με μεταφορά. Όμως, έστω και έτσι συμβάλλει η Γεωργία όσον αφορά τα, τις εκπομπές αυτές και άλλωστε έχουμε τάξει κάποιους στόχους για τη μείωσή τους. Τώρα, τη συμφωνία που θα προκύψει στην ε, Κοπενχάγη θα πληθεί κάποια συμφωνία, οπότε θα πρέπει και εμείς να ανεβάσουμε τον πύχη όσον αφορά τα επιθυμητά επίπεδα των ε, εκπομπών. Άρα θα πρέπει να κάνουμε μια προβληματιστούμε όσον αφορά τις τεχνικές, όσον αφορά τις πρακτικές ε, για τα φαινόμενα του, για τα αέρια του θερμοκηπίου. Το δε βασικό μήνυμα που θέλουμε να προωθηθεί με αυτό το έργο εργασία του φθινοπόρου προς το Συμβουλίο είναι ότι η καλύτερη μέθοδος είναι να έχουμε κάποια μέτρα που συνδυάζουν παραγωγικότητα και βιωσιμότητα. Και έτσι ό,τι και να κάνει κανείς, πηγαίνει κερδισμένος. Έτσι έχουμε μια συνέργεια, περιορισμός των εκπομπών και προσαρμογή. Και παράδειγμα μια τέτοια συμπεριφορά, τάση νοοτροπία είναι αυτό το έγγραφο που αφορά την προστασία του εδάφου. Έτσι μπορούμε να έχουμε λιγότερο διοξίδιο και το θέλω να διευκολύνουμε και τη γεωργία για το μέλλον. Τώρα, όσον αφορά την κοινή αγροτική πολιτική, εμείς σε μια σειρά εγγράφων προσέχουμε τις απόψεις μας. Όπως είναι η ΚΑΠ, έχει συμβάλει στις βλεπτικές εκπομπές. Τώρα, όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, Και έτσι έχουμε βοηθήσει στις, στον υπόλοιπο λίγο της εκπομπής του δύο στον την οδηγία για τα ζωτούχα. Τα, τα μόνιμα βοσκοτόπια και πώς θα προστατευτούν, ε, το δεξιού του άνθρακος και το έδαφος, όλες οι σχετικές προτάσεις μας βοηθούν στην προσαρμογή, στην περιστολή των εκπομπών. Ένα άλλο στοιχείο που αφορά την αρχιτεκτονική της ΚΑΠ είναι το να έχουμε κάποια θετικά κίνητρα στα αντίξιακα προγράμματα τόσο στα κράτη-μέλη και περιφέρειες να μπορούν να διαλέξουν τα μέτρα τα οποία είναι πιο καλά προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους σε σχέση με την προσαρμογή στην ε, αποκατάσταση του κλίματος. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι περιορισμοί, κάποια όρια σε σχέση ας πούμε με την πολλαπλή συμμόρφωση. Άρα αυτή είναι μια προσέγγιση. Η άλλη προσέγγιση είπαμε ότι είναι τα θετικά κίνητρα. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτές τις δύο καθημερινές που μας οδηγούν στα μέτρα για να πετύχουμε το στόχο μας. Και βέβαια θα πρέπει αυτές τις δύο κατευθύνσεις μεταξύ τους να είναι ισορροπημένες. Και τα δύο έρφα τα οποία παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζουν ότι ξέρουμε ποιες είναι οι γενικότερες τάσεις, ξέρουμε τις γενικότερες ε, πτυχές, ξέρουμε ποιες πρακτικές είναι επιβλαβείς και ποιες είναι εποφελείς για τις εκπομπές. Όμως, ακόμα δεν ξέρουμε αρκετά όσον αφορά το τι επιπτώσεις έχει κάθε μας κίνηση, η κάθε μας ενέργεια. Άρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο από πλευρά ακολουθητέων πρακτικών. Και άρα θα πρέπει οι περιφέρειε και τα κράτη-μέλη να κινητοποιήσουν τις, ε, τις ενώσεις των καλλιεργητών. Και θα πρέπει να ε, ενημερωθούν οι γεωργοί με σύμβουλους που θα δράσουν και σε τοπικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Κυρία για τα τόσα σημαντικά που μας αναλύσατε από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βεβαίω και θα συζητηθεί περαιτέρω αυτό το θέμα γιατί είναι τόσο σημαντικό. Γιατί άλλωστε έχουμε και άλλα κοινοβούλια που έχουν ασχοληθεί με το θέμα όπως με το Μεριανικό Συμβούλιο που έχει εμβαθύνει. Έχουν μια κοινοβουλευτική επιτροπή και έχει τις σχετικές πιστώσεις άνθρακα, όπως ονομάζουμε. Θέμα το οποίο πρέπει να ληφθούν υπόψη και σε άλλους τομείς οι οποίοι μολύνουν. Τώρα πάμε τώρα σε άλλο θέμα της διατάξης, το οποίο αφορά την παρουσίαση ενός θέματος συναπόφασης. Για το ίδιο θέμα, Στεφάνη, έχεις το λόγο. Ευχαριστούμε την Κομισιόν. θα πρέπει και εμείς να λάβουμε υπόψη αυτό το οποίο αποφασίστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί έχουμε ας πούμε την ε, Κοπενχάγη και όλες οι κυβερνήσεις πριν από 8 μήνες ε, ενέκριναν μια γραμμή πλεύσης που ενέκρινε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτω ώστε η Ευρώπη να γίνει μοντέλο, πρότυπο για τη μείωση των αερίων, των βλαπτικών για το, για το, θερμοκηπίου. Σε αυτά τα πλαίσια έκαναμε και αυτή την έκθεση. Να μην λαμβάνετε υπόψη ε, κάτι το οποίο βρήκε σύμφωνα στις κυβερνήσει και το κοινοβούλιο είναι λάθος. Το είπε στην αρχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά αυτό το υποπρόγραμμα για το έδαφος, όσον αφορά την ανάλυση για την ε, άνοδο της δημοκρατίας του πλανήτη. Άρα έτσι να πρέπει ως Επιτροπή όχι απλώς να κατεβάσουμε μία γνωμοδότηση, αλλά να κατεβάσουμε μία άποψη. Ευχαριστώ Στεφάνη. Πάρα πολύ εύστοχα αυτά που μας τόνισες. Πριν περάσουμε στο τελευταίο σημείο, που είναι η παρουσίαση τη διαδικασία συναπόφασης προσοχή σε κάτι. Πρέπει να ακούσουμε και πάλι την Κομισιόν, τον κύριο Βεστέιλεν, για ένα αίτημα της Κομισιόν νέα νομοθετική πρόταση για το γάλα. Βέβαια θα έχουμε περισσότερες ειδήσει αργότερα σχετικά με το τι ενέκρινε η Κομισιόν για την κοινή οργάνωση της αγοράς. Αμέσως το λόγο λοιπόν στην Κομισιόν. Κύριος Βεστέιλεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο. Η πρόταση που ενέκρινε η Κομισιόν εγγράφεται μέσα στα άλλα μέτρα που ήδη έχουμε εφαρμόσει για το γάλα και προτάσει που κάναμε στο Συμβούλιο αυτή η πρόταση συγκεκριμένα και ζητούμε επιγόντως να την προσέξετε αποτελείται από δύο μέτρα. Το ένα είναι για την αναδιάρθρωση. Έχουμε νομική βάση στην ενιαία κοινή οργάνωση αγοράς για να αγοράσουμε ποσοστώσεις και να βάλουμε τις ποσοστώσεις αυτές στο απόθεμα και μετά να τις χρησιμοποιούμε για αναδιάρθρωση. Τώρα, προτείνουμε η ποσόστοση που παραμένουν στις 31 Μαρτίου στο αποθεματικό να μην χρησιμοποιούνται για να αντισταθμίσουν να, να δοθούν σε γεωργούς που θα πάνε πέραν των προσωπικών τους ποσοστώσεων. Όπως ξέρετε υπάρχει μια αντιστάθμιση στο τέλος του χρόνου μεταξύ γεωργών που υπερέβησαν τις ποσοστώσεις λαμβάνουμε φυσικά υπόψη και τις ποσότητες στο αποθυματικό και οι ποσότητες αυτές που αγοράζονται για τα προγράμματα αναδιάρθρωσης δεν χρησιμοποιούνται για δύο χρόνια για να δοθούν στα διστάθμισμα σε γεωργούς που υπερβαίνουν τις δικές τους ποσοστώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε μια πληρωμή, έγκυρη πληρωμή υπερισφοράς, super levy, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναδιάρθρωση. Δεύτερο, θα αποθανηθούν οι γεωργοί από το να υπερβαίνουν τις προσωπικές τους ποσοστώσεις. Το δεύτερο μέτρο αφορά τα γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα με βάση το άρθρο 186 ρήτρα διαταραχή που επιτρέπει στην Κομισιόν να λάβει επίγοντα μέτρα στην περίπτωση που υπάρχει διαταραχή. Είδαμε ότι στην τρέχουσα κρίση στα γαλακτοκομικά η Κομισιόν δεν έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της να παρέμβει. Γι' αυτό θέλουμε και το γάλα να συμπεριληφθεί στο άρθρο 186. Να μπορούμε να παρεμβαίνουμε πιο έγκαιρα. Αυτά είναι τα στοιχεία της πρότασής μας και θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν η Επιτροπή σας και το Ευρωκοινοβούλιο γνωμοδοτήσει εγκαίρως έτσι ώστε το Συμβούλιο να μπορεί να πάρει απόφαση για τα μέτρα αυτά το Νοέμβριο ή το αργότερο το Δεκέμβριο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος κάτι για τη διαδικασία. Η Κομισιόν μας ζητάει να γνωμοδοτήσουμε επιγόντως για την νομοθετική αυτή πρόταση. Πρώτο, πρέπει να ορίσουμε την επόμενη Δευτέρα έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, της Γεωργίας, στο Στρασβούργο, για να αποφασίσουμε αν θα δεχτούμε ή όχι αυτό το αίτημα της επίγουσας διαδικασίας. Όπως ξέρετε, το Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια πρέπει να αποφανθεί ναι ή όχι. Την επόμενη Δευτέρα, μετά την Ολομέλεια, έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας για να αποφασίσουμε τι θα πούμε την Τρίτη το πρωί. Δεν υπάρχει λόγος να συζητήσουμε σήμερα η Κομισιόν ανακοίνωσε ορισμένα νομοθετικά μέτρα. Τα εκτιμούμε. Ίσως να υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις στην Επιτροπή μας. Θα τα συζητήσουμε στην έκτακτη συνεδρίαση την επόμενη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Σκεφτείτε το. η συνεδρίαση αυτή θα γίνει ταυτόχρονα με τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών. Και την επόμενη Δευτέρα συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο. Και νομίζω μπορούμε να πούμε εξ ονόματος όλων στην Κομισιόν, περιμένουμε η Κομισιόν να μας εξηγήσει με λεπτομέρειες τι συγκεκριμένα θέλει να κάνει χρησιμοποιώντας το εργαλείο του άρθρου 186. Οι περισσότεροι από εμά θα συμφωνούσαμε να μπει και το γάλα με το κρέας και λοιπά με άλλους τομείς υπό το άρθρο 186. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να ακούσουμε συγκεκριμένα τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν όταν θα της δοθεί αυτή η εξουσία άμεσης παρέμβασης στον τομέα αυτό. χωρίς να χρειάζεται τη γνώμη του Συμβουλίου. Στη συνεδρίαση της Τρίτης, όταν θα γνωμοδοτήσουμε, ας πούμε υπέρ ή κατά για την επίγουσα διαδικασία, να υπάρχει ήδη κάποιος προσανατολισμός εκ μέρους της Κομισιόν πώς συγκεκριμένα σκοπεύει να εφαρμόσει αυτά τα νέα μέτρα. Αν κανείς θέλει να μιλήσει θα του δώσω το λόγο. Αλλά όπως σας είπα, η συζήτησή μας επί της ουσίας θα γίνει τη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Λουίς Καπούλα Σάντος. Πρόεδρε, ξέρω ότι δεν είναι τώρα η ώρα να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Όμω θέλω να υποβάλω μία ερωτησούλα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι υπάρχει μία αντίφαση. Εάν συμφωνούμε όσον αφορά τα πλεονάσματα της προσφοράς, τότε δεν θα πρέπει να αυξάνει την παραγωγή με τα υπολείμματα. Τι θα κάνει για την προσφορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι προτείνει. Γιατί επιμένει σε αυτή την πρόταση εις το να μένουν αμετάβλητε οι αιτήσει ποσοστώσεις. Για μένα αυτό είναι μια αντίφαση. Μένουν σε κάποιο αποθεματικό ε, ε, οι ποσοστώσεις που διατηρούνται, αλλά οι αιτήσει μένουν ίδιες. Αυτό νομίζω ότι είναι, όπως έχει σημαίνει κατάσταση, αντιφατικό. Θέλει άλλο το λόγο, λέει ο πρόεδρος. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι για το ότι τη Δευτέρα θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε αναλυτικά τις προτάσεις Κομισιόν. Δύο πράγματα θέλω να υπενθυμίσω, το είπα προλαλή σας. Πρέπει να υπερασπίσουμε κάποια πράγματα στο κοινό, στους φορολογούμενους και δεν πρέπει βεβαίως από τη μία να λέμε πως αυξήσαμε τις ε, ποσοστώσεις και από την άλλη μεριά και άρα έτσι την προσφορά και μετά να λέμε στα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι πάλι ακριβώς για τις ποσοστώσεις. Δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσουμε αυτό. Και δεύτερον, στην Ανατολική Γερμανία έχουμε σταθερά χαμηλότερες ε, τιμές ε, για την ποσόστοση από ότι στο δυτικό κομμάτι της Γερμανίας. Αυτό κατά βάση οφείλεται στο ότι στα λεγόμενα νέα κρατήδια ε, είχαμε χρησιμοποιήσει αρκετά πάρα πολύ αυτή την λεγόμενη εξυγίανση του τομέα της γεωργίας, κάτι το οποίο επηρεάζει αρνητικά τις ε, τιμές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα δεν θέλω να γίνει συζήτηση ουσίας μόνο το... Ε, επί της διαδικασίας. Συμφωνούμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα την Δευτέρα. Μετά την Τρίτη, όπως είπατε, 9 η ώρα έχουμε την ψηφοφορία στην Ολομέλεια και θα πω το εξή μόνο. Εάν ε, γίνει αποδεκτό, έχουμε την Τρίτη Τετάρτη, με συγχωρείτε, προθεσμία για τις ε, τροπολογίες και πέμπτη ε, έχουμε την ψηφοφορία στην όνομα Απλά το λέω στους συναδέλφους για να μην ε, ζητάει ο καθένας μονομένη εξήγηση. Πρόεδρος, μάλιστα, ο Μάτι Ρόστιν. Επαναλαμβάνω, η συζήτηση θα γίνει τη Δευτέρα του το απόγευμα, το βράδυ, σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, ταυτόχρονα με το Συμβούλιο Υπουργών που θα συνάδει στο Λουξεμβούργο. Μεθοδολογικέ παρατηρήσει σήμερα, επί της ουσίας τη Δευτέρα. Συμφωνώ. Ε, θα θέλαμε κάποιες ε, πληροφορίες, ειδικά για το δεύτερο τμήμα όπου μιλάμε για τις ρήτρες του πώς θα τεθούν αυτά τα πράγματα. Ενισχύει, θυμά, υπενθυμίζω εδώ πέρα πως θα έχει και περισσότερα δικαιώματα όταν τεθεί ενισχύ η λίσαβόνας Λισαβόνα στο Κοινοβούλιο. Οπότε δύσκολο είναι αυτή τη στιγμή να παραχωρήσουμε δικαιώματα. Αυτό θα ήθελα να σκεφτούμε. Αλλιώς, ναι, όπως είπατε, η συζήτηση θα γίνει την Δευτέρα και καλό θα ήταν πριν η συζήτηση να έχουμε τελικά ψηφοφορία. Grazie Martin, Για να δω αν κατάλαβα καλά. Η Κομισιόν μα προτείνει δύο μέτρα. Ένα τεχνικό μέτρο που υπάρχει ήδη στι ποσοστώσεις και το άρθρο 186. Ο Μάρτιν ζήτησε εξηγήσει για το 186. Ένα είναι αυτό. Εγώ παραξενεύομαι όμω, όπως και ο συνάδελφος μίλησε πριν, γιατί μας λέτε τώρα ότι υπάρχουν τεχνικά εργαλεία για να λυθεί το πρόβλημα της παραγωγής, ενώ επί δεν υπήρχαν. Και το Συμβούλιο Υπουργών την περασμένη εβδομάδα δεν μπόρεσε να αναγγείλει τίποτα. Υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα. Εγώ θα ήθελα τη Δευτέρα στη συνεδρίασή μας να έχουμε τα τεχνικά στοιχεία. Μιλήσατε για ένα, υπάρχουν κι άλλα. Τι γίνεται με αυτούς που περνάνε στη σύνταξη, η παραγωγή τους, τι γίνεται. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Το θέμα αυτό το ξέρετε πολύ καλά όλοι σας. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε αν δεν μιλήσουμε για τις νέες ισορροπίες στην Ευρώπη. Σήμερα υπάρχουν χώρες που δεν μπορούν να παράγουν στο ύψος των αναγκών τους. Ε, κυρία Ματιέ, ήθελα εξηγήσει για το άρθρο 186, κύριε Πρόεδρε, εκ μέρου τη Κομισιόν. George Lyon και μετά ο λόγος πάλι στην Κομισιόν. Μία απλή παρατήρηση. Μπορούμε να έχουμε εγγύηση ότι θα έχουμε τις πληροφορίες αυτές το αργότερο μέχρι την Πέμπτη για να, συζητήσουμε, για να μελετήσουμε το θέμα αυτό το Σαββατοκύριακο γιατί ένα που δημιουργεί απογοήτευση είναι ότι δεν έρχεται εγκαίρως πληροφορία στην Επιτροπή μας. Θέλουμε να έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Θα μπορούσαμε να πάρουμε μια απόφαση σήμερα. Μπορούμε να έχουμε εγγύηση ότι θα έχουμε τις πληροφορίες αυτές εγκαίρως, έτσι ώστε Δευτέρα το πρωί να ξέρουμε γιατί αποφασίζουμε. Πρόεδρος διευκρινίζω κάτι για τον Τζόρτζ και για όλου. Στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας τη Δευτέρα στο Στρασβούργο φυσικά θα ζητήσουμε περισσότερε πληροφορίε. Φυσικά δεν μπορεί να έρθει η Επίτροπος γιατί η Φίσσαλ Φίσλαμπερ θα είναι στο Λουξεμβούργο με του υπουργού. Μακάρι να έρθουν οι εκπρόσωποι της Κομισιόν που να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Το ζητάμε ήδη από τώρα αυτό. Όχι σήμερα. Σήμερα κάτι μεν, αλλά θα γράψω επιστολή στην Επίτροπο για περισσότερες λεπτομέρειες τη Δευτέρα. Για το 186, οπωσδήποτε για τη συνάδελφα Ματιέ, πρέπει η Κομισιόν να δώσει απάντηση. Κομισιόν. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα. Θα απαντήσω να είμαι σαφής. Υπάρχει νομική βάση στην ε, ενιαία κόα για να εξαγοραστεί πόσο είναι το άρθρο 75 και μέχρι τώρα οι ποσότητες που ήταν στο απόθεμα π.χ. στις 31 ε, Μαρτίου όταν ξεκινάμε την αξιολόγηση την υπέρβαση της ποσόστοσης ελήφθησαν υπόψη για να αποσμειωθούν οι αγρότες. Η πρόταση είναι τώρα να μην χρησιμοποιηθούν αυτές οι ποσότητες, οπότε το μέσο αναδιάρθρωσης υπήρχε πάντα. Και το πλεονέκτημα είναι πως υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες οι αγρότες θα πληρώνουν ε, πάρα πολλά, ένα επιπλέον τέλος σε κάποια αρχική φάση που θα χρησιμοποιηθεί μετά για να διαρθρωθεί. Τώρα, όσον αφορά το άρθρο 186, εξαρτάται βεβαίως από το τι είδους κρίση έχουμε και τι μέτρα μπορούμε να λάβουμε. Αλλά, παραδείγματος χάνει προς στιγμή δεν έχουμε νομική βάση για ιδιωτική αποθεματοποίηση διαφόρων προϊόντων πλην βουτύρου στον ενιαία, στην ενιαία ΚΟΑ. Οπότε σε μια μελλοντική κρίση η ιδιωτική αποθεματοποίηση μπορεί να, να χρησιμοποιηθεί. Οπότε αυτό είναι ένα παράδειγμα χρήση του άρθρου 186. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπε η Κομισιόν. Εύχομαι στην έκθεση που θα μας κάνετε στη Γενική Διεύθυνση, η Γενική Διεύθυνση, να καλυφθεί το ενδιαφέρον της Επιτροπής μας. ότι αυτό που ψήφισε το Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια με μεγάλη πλειοψηφία και για την νομοθετική πρόταση και για το ψήφισμά μας που το ψήφισαν πάνω από 450 βολευτές να ληφθεί υπόψη από την Κομισιόν. Το 186 μας λέτε είναι ένα εργαλείο που μπορεί να επιτρέψει να ληφθεί υπόψη αυτό που ζήτησε το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Θα τα συζητήσουμε στη συνεδρίασή μας τη Δευτέρα το βράδυ. Και φυσικά ελπίζουμε να είναι παρούσα η Κομισιόν. Και τώρα περνάμε στο επόμενο και τελευταίο σημείο της ε, ημίρησης διάταξης, παρουσίαση της διαδικασίας συναπόφασης πολύ σημαντικό θέμα διδακτικού χαρακτήρα. Μετά την ψήφο της Ιρλανδίας και χάρη στο σημαντικό αυτό αποτέλεσμα έχουμε τώρα την εφαρμογή της συναπόφασης ελπίζοντας ότι ο τελευταίος ύφολος μετά την καλή είδηση του περασμένου Σαββάτου που ότι υπέγραψε ο Πολωνός Πρόεδρος τη συνθήκη της Λισαβόνας Τώρα μένει ένας τελευταίος ύφαλος. υπογραφή εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τσεχίας. Αλλά ήδη αρχίζουμε και ετοιμαζόμαστε για το σημαντικό αυτό ραντεβού. Για να ξέρουμε λοιπόν τι σημαίνει για την Επιτροπή μας η επίσημη εφαρμογή της συναπόφασης, πρέπει όλοι να προσέξουν, να δώσουμε προσοχή στην τεράστια σημασία που θα έχει η συναπόφαση για τις επιλογές μας. Γι' αυτό ζήτησα από τον υπεύθυνο για την διαβούλευση συναπόφαση από τη γραμματεία του γραμματείου, από τον κύριο Κλάους Μπάιερ, να μας κάνει μια σύντομη εισαγωγή. Όπως βλέπετε, μοιράζουμε το μικρό αυτό φυλάδιο, πάρα πολύ σημαντικό, σε όλες τις γλώσσες ή τουλάχιστον στις περισσότερες γλώσσες της Ένωσης για να ξέρετε εγκαίρως τις νέες σημαντικές εξουσίες που θα έχει και η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας. Ο κύριος Κλάους Μπάγερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μου δίνει ευκαιρία σήμερα να απευθυνθώ στην Επιτροπή Γεωργίας και σύντομα να σας παρουσιάσω τη διαδικασία της συναπόφασης. Κατά εκταντήρηση να συνεχίσω επαναλαμβάνοντας τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της διαδικασίας και στη συνέχεια να δούμε τι θα αλλάξει με την συνθήκη της Λισαβόνας. Ελπίζουμε σύντομα να τεθεί σε ισχύ. Ήδη ο Πρόεδρος ανέφερε αυτό το φυλάδιο το οποίο έχει διανεμηθεί και εκεί σε σύνοψη εκθέτουμε Ποια είναι η διαδικασία στο Κοινοβούλιο, αλλά επίση ε, κοιτάξτε και το παράρτημα, διότι εκεί πέρα υπάρχουν διάφορα χρήσιμα έγγραφα, όπω άρθρα τη συνθήκη, ε, διαδικαστικά, κανονών κώδικα διοντολογία κλπ. Τώρα, μία μικρή εισαγωγή. Ε, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της διαδικασίας. Η διαδικασία της συναπόφαση μόνη νομοθετή διαδικασία για Κοινοβούλιο και Συμβούλιο όπου ενεργούν σε ισότητα. Το 1993 με στιγμή του Μαστρίχτ ε, ξεκίνησε αυτή η ιστορία και αφορά μισές πολιτικές ένωσης. Προβλέπονται τρεις αναγνώσεις. Όμως προβλέπεται ότι είναι δυνατόν και σε μία αναγνώση να κλείσει το θέμα Είτε στην πρώτη, στην στην τρίτη. Και πάρα πολλές φορές ισχύει και τέτοιο, δηλαδή ε, κλείνει κάθε φάκελο, στο κάθε θέμα νωρίς στην πρώτη ανάγνωση. Διαφορετική κανόνε κίνηση στην πρώτη φάση, διαφορετική στη δεύτερη, διαφορετική στην ε, συνδιαλλαγή. Βασικές διαφορές για να τα πούμε δύο λόγια, είναι ότι στην πρώτη ανάγνωση δεν έχουμε προθεσμίες. Άρα προετοιμάζονται τα θεσμικά όργανα, όμως οι βασικές διαφορές μεταξύ πρώτης και δεύτερης ανάγνωσης είναι ότι στη δεύτερη ανάγνωση το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει μια απόλυτη πλειοψηφία. 369 βουλευτέ, δηλαδή θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ κάποια συγκεκριμένη τροπολογία. Άρα, το κατόφλι δεύτερη ανάγνωση είναι πολύ ψηλότερο από ό,τι στην πρώτη αναγνωσή. Μια άλλη διαφορά τώρα είναι υπό ποιους όρους είναι μια τροπολογία αποδεκτή. Στη δεύτερη ανάγνωση το Κοινοβούλιο περιορίζεται από το τι τροπολογίες θα υποβάλει, ε, περιορίζεται από τον ίδιο του τον κανονισμό. Πολύ σύντομα. Προαναφέραμε ότι είναι πολύ διαφορετική από την πρώτη δεύτερη ανάγνωση η τρίτη ανάγνωση. Διότι στην τρίτη ανάγνωση προβλέπει η συνθήκη τη διαδικασία της συνδιαλλαγής. Είναι κάτι σαν τελευταία ευκαιρία να επιτευχθεί συμφωνία. Εάν δεν έχει επιτευχθεί προηγουμένω. Προβλέπεται η συνάντηση, η συνεδρίαση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής. Έχουμε την αντιπροσωπεία του Συμβουλίου και την προσωπία του Κοινοβουλίου. Συναντιούνται και προσπαθούν να τα βρουν. Και αυτό γίνεται μόνο στην τρίτη ανάγνωση. Μόνο τότε έχουμε τέτοια συνάντηση. Έχετε εδώ πέρα μια ανάλυση του πώς χρησιμοποιούνται αυτές τις διαδικασίες σήμερα. Βλέπετε και εδώ στην οθόνη και η τελευταία στήλη είναι η τελευταία ε, θητεία, 2009. Εκεί βλέπετε ότι περισσότερο από δύο, δύο τρίτα των θεμάτων κλείσανε στην πρώτη ανάγνωση. Κάτω από 30% πήγε στην συνδιαλλαγή. Αλλά τα περισσότερα πήγανε σε πρώτη ανάγνωση. Για κοιτάξτε τι έγινε στις προηγούμενες δύο όμως ε, θητείες. Θα δείτε ότι υπάρχει μια βασική τάση. Όλα είναι υπόσταση είναι στην πρώτη ανάγνωση. Και αυτό γιατί γίνεται, διότι τα θεσμικά όργανα τώρα εμπιστεύονται τον το άλλο περισσότερο και συνομιλούν ούτως υπήν νωρίτερα, καλύτερα, περισσότερο και επίσης ε, υπάρχει πολύ καλύτερη εξοικείωση όλων με αυτή τη διαδικασία. Το βασικό πλεονέκτημα τώρα είναι ότι έτσι εξοικονομείται χρόνος και η διάρκεια είναι 6 μήνες από την υποβολή της πρώτας κομισιόν μέχρι την δημοσίευση στην εφημερίδα την επίσημη. Και αυτό είναι σύντομη περίοδος, ακόμα και για εθνική νομοθεσία και είναι ιδιαίτερα σύντομο. Αλλά δημόσια το πρέπει κινούμεθα σε περιβάλλον πολυγλωσσίας. Και άρα η πρώτη κομισιόν, η τροπολογία το ελληνικό κείμενο, όλα μεταφράζονται σε όλε τι γλώσσε. Και όλα αυτά ολοκληρώνονται σε 16, όχι 6 μήνε. Είδα τώρα τι έγινε, ιδίω στο δεύτερο ήμιση τη τελευταία θητεία. Εδώ στο Κοινοβούλιο είχαμε πάρα πολλέ επικρίσει οι οποίε ακούστηκαν για τις σημαίες που επιτεύχθηκαν στην ε, πρώτη αναγνώριση και είπαν ότι δεν χαρακτηρίζονται από εκεί πάρα πολύ μεγάλη διαφάνεια και αυτοί που παρακολουθούν τις εξελίξεις είπαν ότι δεν μπορούν να τις παρακολουθήσουν. Το πώς κλείνονται τα θέματα, εάν τα θέματα κλείνουν τόσο νωρί. Επίση και τα Εθνικά Κοινοβούλια παραπονέθηκαν αρκετά και μα είπαν ότι πάρα πολύ δύσκολο είναι να μπορούν να ασκήσουν κοινοβουλευτικό έλεγχο προ την εθνική του κυβέρνηση εάν έχουμε το, το τόσο μεγάλο τμήμα, 72% δηλαδή των θεμάτων που κλείνουν τόσο νωρί Γι' αυτό και το 2007 έχουμε μια ομάδα εργασία που συγκροτήθηκε στο Κοινοβούλιο. Επικεφαλής τέθηκε η κυρία Ροτ Πέρεντ. Εξετάστηκε που μπορεί να βελτιωθεί στην απόφαση. Η δε ομάδα αυτή εργασίας πρότεινε ένα κώδικα δεοντολογίας για να γίνεται η διαπραγμάτευση σε πρώτη και δεύτερη ανάγνωση. Και έτσι, αυτός ο κώδικας δεοντολογίας ενσωματώθηκε στο κοινωνισμό του Κοινοβουλίου. Αυτός, ο οποίο τον Ιούλιο άρχισε να ισχύει. Εδώ και μόλι λίγο είναι πολύ φρέσκο αυτό το έγγραφο, να σα πω δύο λόγια βασικός στόχος αυτού του κώδικα είναι να έχουμε περισσότερη διαφάνεια στη διαδικασία. Το πνεύμα που διαπνέει αυτή τη εργασία είναι το ότι θα έχουμε περισσότερη διαφάνεια. Εάν ο τριγωνικός διάλογος συνδέεται πάρα πολύ με την πηγή, με το σώμα που από ξεκίνησε το Ρεβαδέλη δηλαδή Κοινοβουλική Επιτροπή. Αν δηλαδή ας πούμε για ένα γεωργικό θέμα ενημερώνεστε εσείς. Και έτσι έχουμε περισσότερη διαφάνεια και ενημερώνεται και το κοινό. Και η Γενοστική Επιτροπή πρώτα απ' θα αποφασίσει για τις διαπραγματεύσεις. Θα αποφασίσει ποιος θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις. Ίσως ο συγητής και οι σκιώδε. Ποιος θα είναι στην επανειληπτική ομάδα. αποφασίζει η Επιτροπή την ε, διαπραγματευτική εντολή και υπάρχει και feedback προς αυτήν από τους διαπραγματευτές τώρα. Έτσι παρακολουθεί καλύτερα και ο κόσμος το νομοθετικό έργο. Υπάρχουν περισσότερες εγγύσεις προς τούτο. Ενημερωτικά σας παραμένω σε αυτό το εγχειρίδιο, αυτό το βιβλιαράκι, μπορείτε να βρείτε τον κώδικα για στο παράδειγμα Δέλτα. Τώρα, πριν έρθουμε στα της Λισαβόνας, να σου δώσω κάποια στοιχεία από την τελευταία θητεία. Συνολικά. Είχαμε 453 454 θέματα τα οποία κλειστήκαν από τη συνδιαλογή. Βλέπετε εδώ πέρα είναι η κατανομή σε σχέση με τις ε, κοινωνικές επιτροπές. Envy 20%, Γιούρι 18%, Τραν 11%, Οικονομική 8%, είχατε διατροφική ασφάλεια και στατιστικά. Όμω, η υποστήριξη τη Λαβάνα σε πέντε χρόνια τελείω διαφορετική θα είναι η κατανομή τη πίτα. βρισκεί η συνήθεια τη Λισαβόνα και μια από τώρα τι θα αλλάξει η συνήθεια τη Λισαβόνα όσον αφορά την νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Πρώτα-πρώτα, δεν θα έχουμε απόφαση. Θα έχουμε μια συνήθεια νομοθετική διαδικασία όπως το ονομάζεται. Και το κείμενο της σχετικής συνθήκης ε, ξαναδιατυπώθηκε ούτω ώστε να μπορούμε να είμαστε σε ισότιμο το Κοινοβούλιο. Δεν μιλάει για γνώμη, μιλάει για θέση του Κοινοβουλίου. Η διαδικασία δεν είναι στην ουσία της. Έχουμε πάλι τρεις αναγνώσεις και τις ίδιες προθεσμίες. Όμως βέβαια εδώ αλλάζουν κάπως οι, οι εμπλεκόμενοι. Έχουμε τον έλεγχο της επικουρικότητας. Και στο μέλλον θα έχει το κοινοβούλιο 8 εβδομάδες για να μπορέσει να αντιδράσει η πρόταση της Κομισιόν. Εάν θεωρούν ότι η πρόταση της Κομισιόν δεν είναι σύντονη με την επικουρικότητα. και ανάλογα με το τι θα πούν τα Εθνικά Κοινοβούλια υπάρχουν διαφορετικές παραγές διαδικασίας, Α ε, ας πούμε κίτρινη κάρτα κλπ. Η κόκκινη κάρτα. Και εάν το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο ακολουθεί τη γνώμη του ότι δεν, ε, δεν, γίνεται, δεν, δεν τηρεί την τότε σταματάει η διεκπαιρέωση του θέματος. Μια άλλη διαφορά τώρα η οποία πάρα πολύ σχετίζεται με την συναπόφαση, είναι το όρο καθεστώς της επιτροπολογίας. Το πώς της πίζονται κάποια μέτρα. Η ιεράρχηση κανόνων προβλέπεται από τη στιγμή της Λισαβόνας, σε σχέση με νομοθετικές πράξεις, που τώρα θεσπίζονται είναι και η κατανάθεση πράξη από μια μεριά, ενώ είναι εφαρμοστικέ πράξεις. Η κατανάθεση πράξης είναι οι πιο αυστηροί να σας πούμε, δηλαδή ότι έχουμε τους συνομοθέτες, ονειοβούλιο και συμβούλιο, που αναθέτουν κάποια μέτρα να τα λάβει η, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως ταυτόχρονα διατηρούν τα δικαίωμα της κυρίας, για να διαφωνούν με την πρόταση. Τώρα, οι εφαρμοστικές πράξεις, αυτά είναι τα πιο λεπτομερή νομοθετήματα, είναι πράξεις που ανατίθενται στα κράτη-μέλη. Όμως, η Κομισιόν όταν χρειάζεται ομοιομορφία μπορεί εκείνη να θεσπίσει κάποια μέτρα. Τώρα στον αφορά το όλο πλαίσιο θα πρέπει να εγκριθεί από τα τρία θεσμικά όργανα. Η πιο σημαντική όμως αλλαγή είναι η εμβέλεια της συναπόφασης στο μέλλον. Όλες οι βασικές πολιτικές θα διέπονται από αυτή τη διαδικασία με εξαίρεση κάποιες πάρα πολύ λεπτές ε, πολιτικές όπως φορολογική πολιτική, πολιτική ασφάλειας, κάποιες, ε, κάποια παρακάτες της κοινωνικής πολιτικής, οπότε έχουμε 85 αντί για 44 τομείς που καλύπτονται τώρα. Και μπορείτε να βρείτε ένα κατάλογο από όλα αυτά εδώ στο φυλάδιο αυτό. Τώρα για, για το κοινοβούλιο σημαίνει αυτό ότι θα έχουμε τέσσερις κοινοβουλικές επιτροπές που θα έχουν πάρα πολύ δουλειά λόγω της συναπόφασης. Πρώτα πρώτα δική σας επιτροπή, η Επιτροπή Γεωργίας, αλλά και η Επιτροπή Ελίας. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου επίσης, αλλά και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Οπότε μπορώ εγώ παρά να σε ευχηθώ. Καλή επιτυχία. Καλό κοράγιο. Και ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Κλάς της Γενικής Γραμματείας. Μελετήστε όλοι σας το βιβλιαράκι αυτό, είναι πολύ έτοιμο. κλείνει η συνεδρίαση της Επιτροπής. Σας θυμίζω τη συνεδρίαση την επόμενη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Έκτακτη συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίαση 9 και 10 Νοεμβρίου. Πέρα συνεδρίασης 5 λεπτά διακοπή και παρακαλώ να μείνουν οι Μετά.